Je vous propose que nous commencions... Euh, Καλημέρα. Να αρχίσουμε απευθείας την ε, σημερινή μας ακρόαση για τα προβλήματα κοινωνικής ένταξης των γυναικών που ανήκουν σε εθνικές μειονοτικές ομάδες. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους και όλες. Προφανώς ε, θα ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Αντώνια Παρβάνοβα, η οποία είναι η συγγήτρια μας ε, για τους ε, μετανάστες και τις εθνικές μειονοτικές ομάδες και ευχαριστώ εκ των προτέρων τους εμπειρογνώμονές μας που θα καταθέσουν τη μαρτυρία τους, τις εμπειρίες τους, στη σημερινή μας ακρόαση, θα είναι στη διάθεσή μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Η κυρία Γκράινερ που είναι η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Μεταναστριών στη Γερμανία, η κυρία Ιζαμπέλα Νικαλάκη, αναπληρώτρια διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των ρωμ Θα κάνετε τις πρώτες παρεμβάσεις στη σημερινή μας συζήτηση. Ο κύριος Φωτάκης, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα παρέμβει στην ακρόασή μας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Κατόπιν θα κάνουμε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συζητήσεις για τις πρακτικές ως προς την ένταξη με την κυρία Μέλλερ Γένσεν από το Δανικό Κέντρο Ενημέρωσης για τις γυναίκες και την ισότητα των δύο Φίλων και φυσικά τον κύριο Εγιούπ, πρόεδρο της Επιτροπής για την Προστασία κατά της διακριτικής μεταχείρισης της Βουλγαρίας. Καλώς ορίσατε. Στο τέλος του πρωινού θα έχουμε και άλλες παρεμβάσεις ε, από την κυρία Μπαχ, από το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών, παραδείγματο χάρη, που θα μας κάνει κάποιες εισηγήσεις. Σας ευχαριστώ όλους και θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα. Ε, και θα ε, καθυστερήσει, θα ε, φύγει σε λίγο, συγγνώμη, για να πάει να ψηφίσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Παρακαλώ, στο μεταξύ σας ακούμε. Thank you, uh, Mrs. Maureen uh, Chartier, dear colleague. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, τη συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που είμαι εδώ σήμερα και συζητάμε το σημαντικό το θέμα της κοινωνικής ένταξης των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων από πρώτα απ' όλα πως η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φίλων ε, αποδίδει μεγάλη σημασία σε αυτό το ζήτημα και βεβαίως ε, θα καλωσορίζουμε την ακρόαση αυτή και θα ακολουθήσει μια έκθεση και βεβαίως ε, θα συζητήσουμε και τα προβλήματα γυναικών που ανήκουν σε γνωστές ομάδες μειονοτήτων και σε αυτές που ανήκουν σε μεταναστευτικές κοινότητες. Είναι φιλόδοξος ο στόχος, αλλά θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων να δούμε τις διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων και να δούμε αν υπάρχουν διαφορές ε, σε κάποιες ε, διακριτικές μεταχειρήσει ε, εις γυναικών που ανήκουν σε μειονότητες ή είναι μετανάστες μέλος της Επιτροπής και η συγητής, συγητρία. Και όπως ε, όλοι οι βουλευτές ε, δίνουμε μεγάλη σημασία σε εκθέσεις που δημιουργούν το πολιτικό και νομικό περιβάλλον, δεδομένου ότι ζούμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία που συμπεριλαμβάνει πολλές ε, Διακριτές ε, θρησκευτικές ε, πολιτιστικές ε, κοινότητες. Πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα αυτό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τονίσουμε το ότι το να είναι κάποιος γυναίκα που ανήκει σε μια εθνοτική ομάδα δεν είναι αναπηρία σε μια δημοκρατική κοινωνία, αλλά παίζει ένα σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό ρόλο. Οπότε το αντικείμενο της έκθεσής μου θα είναι να αξιολογήσουμε τις σχετικές πολιτικές της Ένωσης για ενσωμάτω... στην Ένωση για ενσωμάτωση γυναικών που ανήκουν σε μειονότητες και να δούμε ποιες είναι οι λύσεις. Ε, τα δύσκολα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να δω είναι ο ρόλος των πολιτικών σωμάτων, ο ρόλος των γυναικών και της ε, πολιτικής ισότητας ε, των φίλων για να υπάρξει αποτελεσματική ενσωμάτωση καθώς καμιά φορά οι ανάγκες είναι συγκρουόμενες θα πρέπει αυτές να συμβαστούν οπότε θα πρέπει να δούμε αυτές τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και να βρεθεί ένας τρόπος να συμβιβαστούν για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν οι νόμιμες ε, απαιτήσει αυτών των γυναικών χωρίς βεβαίω να χαθεί η ταυτότητα της εθνικής ομάδας. Δεν υπάρχει μια νομικά δεσμευτική πολιτική της Ένωσης για αυτό το θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως γιατί βεβαίως είναι μια ε, ευθύνη των ε, κρατών μελών. Όμως η πολιτική ενσωμάτωση γίνεται όλο και πιο σημαντική στο επίπεδο της Ένωσης και υπάρχει μια προσπάθεια ενός ε, κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου η Κομισιόν τονίζει πως η ενσωμάτωση γίνεται ακόμη πιο σημαντική με βάση και τη δημογραφική με πτυχή της γύρανσης του πληθυσμού και οι γυναίκε των μειονοτήτων αποτελούν ένα στόχο των πολιτικών ενσωμάτωση. Υπάρχει λοιπόν ο στόχος του να δημιουργηθεί συμμετοχή, να υπάρξει πρόσβαση, να νιώσουν αυτές οι γυναίκε ότι ανήκουν και δεν θα πρέπει να περιοριστούν μόνο σε νομοθετικά μέσα αλλά και σε διοικητικέ και εθελοντικές δραστηριότητες. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω εδώ πέρα κάποιες συνθήκες ε, και παράγοντες που εμποδίζουν την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών από εθνοτικές ε, μειονότητες ε, σε σχέση με τις γυναίκες που ανήκουν στην πλειοψηφία. Έχουμε πρώτα απ' όλα το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, εκπαίδευσης, τη στέγαση και τις δυνατότητες ευρεσής εργασίας. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε τις προσπάθειες και σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο για την πλήρη χρήση των υπαρχών των μέσων και μελλοντικά μέσα για να υπάρξει ενσωμάτωση των γυναικών από εθνικέ μειονότητε για να είμαστε επιτυχεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη. Είμαι εισηγήτρια μιας, έκθεσης, ε, μιας άλλης έκθεσης που θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, οπότε θα φύγω τώρα και θα ξαναέρθω σε λίγο. Σας ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστούμε κύριε Παρβάνοβα για την ε, ταχύτατη ομολογουμένους παρουσίασή σας σχετικά με τους άξονες ε, των ε, σημερινών μας εργασιών. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, στην Επιτροπή μας ε, που δείχνει ιδιαίτερη αφουσίωση για αυτά τα θέματα, για την ισότητα δηλαδή των δύο φύλων ε, σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Εύα Σβένσον, η πρόεδρος μας, έχει κάποιο κόλλημα και δεν θα παρευρεθεί στη σημερινή ακρόαση. Παρόλα αυτά, καταδεικνύει ισχυρή πολιτική βούληση και παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι εργασίε τη Επιτροπή μα. Θα ακούσουμε τώρα τι ευρωγνώμονες. Η κυρία Γκράινερ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταναστριών στη Γερμανία, θα πάρει πρώτη το λόγο. Έχετε 15 λεπτά χρόνο αγόρευσης και θα μεριμνήσουμε ώστε να τηρήσετε αυτό το χρόνο. Παρακαλώ, σας ακούμε. Um, honorable Αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να ε, μιλήσω για ένα ιδιαίτερα προσφυλές για το ευρωπαϊκό μας ε, κέντρο θέμα. Σήμερα εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Μεταναστριών. Εκπροσωπούμε οργανώσεις ε, από διάφορες ε, χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα από διάφορες χώρες, 20 ε, συγκεκριμένα και έχουμε ένα ευρύτατο φάσμα πραγματογνωμοσύνης για όλα τα ζητήματα που άπτονται των μεταναστριών και ασχολούμαστε με θέματα σε εθνικό επίπεδο και ο στόχος μας είναι να συγχρονίσουμε όλες τις εθνικές προσπάθειες και να ε, θεσπίσουμε δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ιδρύθηκε το κέντρο σε μια διάσκεψη που διοργανώθηκε το 2007 στις Βρυξέλλες. Είχαν προσκληθεί διάφοροι εμπειρογνώμονες από διάφορες χώρες για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους ε, ως μετανάστριες ανά την Ευρώπη. Μετά από αυτή την πρώτη συνεδρίαση εκπονήθηκε ένα έγγραφο που ε, τίτλοφορεί το «Ίσα δικαιώματα ε, μετανάστρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Για την κοινωνική ένταξη των ενταναστριών εντοπίσαμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και συνιστούν φραγμούς. Το, η νομική υπόσταση που παρεμποδίζει την κοινωνική ένταξη. Παραδείγματος χάρη όταν κάποιος παντρεύεται με μία άλλο δαπή πρέπει εκείνη να παραμείνει δύο χρόνια στη χώρα πριν να αποκτήσει μόνιμη άδεια παραμονής, παρότι ορισμένε φορές υπάρχει οικογενειακή βία και δυσκολεύονται οι γυναίκες να διαφύγουν από αυτή την κατάσταση. Επίσης, εκπαίδευση και απασχόληση. Τα προσόντα που έχουν αυτές οι γυναίκες είναι ίσα ε, με τον υπηκό της χώρας παρόλα αυτά χρειάζεται να καταβάλουν ε, ιδιαίτερες προσπάθειες ε, στη νέα αυτή χώρα διοργανώνονται πολιτικές εκστρατείες, ε, γίνεται λόμπινγκ, ασκείται πίεση, ούτω ώστε να δούμε πώς ακριβώς, ε, ποιες προσαρμογές μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε τα δικαιώματα αυτών των γυναικών. Επίσης, εργάζονται σε χαμηλόμιστες ε, θέσεις εργασίας αυτές οι γυναίκες, σε υποχείριστες συνθήκες. Επίσης, σεξουαλική υγεία και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Ορισμένες φορές ζουν σε τέτοιες καταστάσεις που δυσκολεύουν Οπότε οι γυναίκες διότι παραδείγματος χάρη δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση ή δεν μπορούν να αποφασίσουν μόνες τους αν θέλουν να ιδρύσουν μια οικογένεια ή όχι. Η ε, βία τώρα κατά των ε, μεταναστριών, ακροτηριασμό των γυναικείων ε, γεννητικών οργάνων, φόνη τιμής, εμπορία γυναικών, καταναγκαστική γάμη, οικογενειακή βία. Για το νομικό καθεστώς θα προτείναμε τα εξής. Να έχουν τις, ε, τη δυνατότητα να έχουν μόνιμες άδειες παραμονής, να έχουν ένα μόνιμο, μια νόμι, νομι, ε, μονιμη νομική υπόσταση στη νέα ε, χώρα τους για όσες γυναίκες δεν έχουν χαρτιά, δεν, έχουν, δεν διαμένουν μόνιμα σε κάποια χώρα και Ορισμένες γυναίκες δεν υπάρχουν νομικός πώς στην κοινωνία και άρα αυτό οδηγεί σε κατάχρηση γιατί δεν μπορούν να πάνε στην αστυνομία, να κάνουν καταγγελίες και σχηματίζουν εξαιρετικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οπότε προτείνουμε πλήρη πρόσβαση στα βασικά δικαιώματα και ανάπτυξη νομικών διάβλων για την νομιμοποίησή τους. Σχετικά τώρα με το ότι δεν αναγνωρίζονται κάποια πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους, θα προτείναμε να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση στον τομέα αυτό. Ε, σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων τους, ε, θα θέλαμε να επιτύχουμε ταχείες ε, διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Επίσης, έχουν περιορισμένες δυνατότητες για περαιτέρω εκπαίδευση, κυρίως επαγγελματικά μαθήματα για συγκεκριμένες ομάδες μεταναστριών. Θα θέλαμε να, προαχθούν, να προαχθεί η επαγγελματική κατάρτιση για αυτές τις γυναίκες. Επίσης, δωρεάν μαθήματα γλωσσών, όχι ομοιόμορφα για ε, όλες τις γυναίκες. Πρέπει να εξετάσουμε ποια προσόντα ήδη έχουν, ε, ούτως ώστε να προσαρμόσουμε τα μαθήματα που προσφέρουμε. σχετικά πάλι με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Ε, ε, υπάρχει περιορισμένη υποστήριξη για τις γυναίκες επιχειρηματίες. Ε, επιθυμούν να στήσουν μια επιχείρηση, αλλά δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς. Πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Επίσης, στο χώρο εργασίας διαπιστώνουμε ισχυρή διακριτική μεταχείριση και πολύ συχνά, παρότι είναι σε χαμηλόμιστες θέσεις εργασίας αυτές οι γυναίκες, ποτέ δεν προάγονται. Ε, Θα βοηθούσε λοιπόν να δημιουργήσουμε ε, ίσες ευκαιρίες για αυτές τις γυναίκες. Ε, τώρα, ε, ευρεία μη ρυθμισμένη απασχόληση. Τι προτείνουμε να εφαρμοστούν οι κανονισμοί σχετικά με την έκδοση αδειών εργασίας. Τώρα, εκμετάλλευση των εργαζομένων που δεν έχουν διαμένουν νόμιμα σε κάποια χώρα. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση στις χώρες εργασίας, κυρίως όταν μιλάμε για χαμηλόμιστες θέσεις θέσει απασχόληση ή θέσει για χαμηλά προσόντα. Ε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προωθήσουμε την ε, ε, επαγγελματική κινητικότητα. Επίσης, ως προς την, υγεία την σεξουαλική υγεία και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα, θα πρέπει να συνεχίσουμε να διοργανώνουμε ενημερωτικές εκστρατείες. Σας μίλησα πριν για τον ακροτηριασμό των γεννητικών οργάνων και άλλες τέτοιες πρακτικές ε, η απόκτηση άλλων γνώσεων θα βοηθήσει πάρα πολύ γιατί υπάρχει ένα χάσμα ενημέρωσης και ως εκ τούτου υπάρχει και έλλειψη κατανόησης των αναγκών τους. Όταν φεύγουν αυτές οι γυναίκες από τις χώρες τους, φέρουν μαζί τους ε, τον πολιτισμό τους, την αντίληψη που έχουν για την αναπαραγωγική υγεία και άρα ε, θα προτείναμε να αναπτύξουμε νέα εργαλεία ως προς την υγεία των μεταναστριών ε, που θα χρειάζονται υπάροχοι κοινωνική κοινωνικής ασφάλισης στις νέες χώρες για να τις καταλάβουν και νέα διεύρυνση των κριτηρίων, τόσο ώστε να δικαιούνται πρόσβαση στα συστήματα υγείας. Τώρα ως προς τη βία, μην ξεχνάμε ότι ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε ειδική νομοθεσία γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο στους ε, εθνικούς ε, φορείς ούτως ώστε να επιτύχουμε μια μηδενική ανοχή για την οικογενειακή βία. Επίσης να προσκαλούμε εμπειρογνώμονες από τις κοινότητες των μεταναστριών για να τις καταλάβουμε καλύτερα και θα προτείναμε να έχουμε συγκεκριμένα μαθήματα εκπαιδευτικά για τους παρόχους υπηρεσιών. Ε, τώρα για την ε, ε, συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έλλειψη γνώσεων για τα πολιτικά συστήματα των χωρών αυτών των γυναικών ως προς την νομοθεσία, τα δικαιώματα ψήφου. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές ανάμεσα στη χώρα καταγωγής και τη χώρα προορισμού. Σε πολλές χώρες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αυτές οι γυναίκες και εφόσον δεν μπορούν να συμμετάσχουν δύσκολα μπορούν να αισθανθούν ότι εντάσσονται σε ένα κοινωνικό σύνολο. Άρα ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η διεύρυνση της συμμετοχής τους και η θα χρειαστεί να αναθέσουμε μεγαλύτερες εξουσίες ε, ε, στις ηγέτιδες αυτών των κοινωνικών ομάδων για να μπορέσουν να προωθήσουν τα δικαιώματα των υπολείπων γυναικών και φυσικά υπάρχει έλλειψη μέσων ε, για τις, για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που ε, παρέχουν αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ως προς τα πολιτικά δικαιώματα αυτών των γυναικών και ε, τελική, τελευταία έλλειψη είναι ότι δεν υπάρχουν κοινωνικά πρότυπα για την συμμετοχή στα κοινά στην πολιτική ζωή. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει το mainstreaming, η ένταξη αυτής της διάστασης ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις μεταναστευτικές πολιτικές σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για να αναγνωρίσουμε τις ειδικές ανάγκες αυτών των μεταναστριών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που δείξατε ε, και στην ε, ιστοσελίδα www.migrantwomen.org θα έχετε σύντομα αυτήν την ε, παρουσίαση που μόλις ακούσατε. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκράινερ για αυτή την σύντομη παρουσίαση. Θέσατε τα προβλήματα που υπάρχουν, ταυτόχρονα δε καταθέσατε και κάποιες ιδέες που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ούτω ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τώρα θα ακούσουμε την κυρία Ιζαμπέλα Μάλκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο των Δικαιωμάτων των Γυναικών ΡΟΜ. Από το 96. δραστηριοποιείται ιδιαίτερα αυτό το κέντρο για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης. Θα σας ακούσουμε με προσοχή, παρουσιάστε μας τις εμπειρίες σας και τη δράση του Ευρωπαϊκού αυτού κέντρου. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Πρώτα απ' όλα να πω και εγώ πως αντικαθιστώ την συναδελφό μου που είναι συντονιστής φίλου και ίσων δικαιωμάτων. Ούτως ή άλλως ε, δούλευα με το σχετικό Ινστιτούτο τα τελευταία 6 χρόνια για αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα λοιπόν να ξεκινήσω με την έλλειψη δεδομένων. Έπρεπε να σκεφτώ πάρα πολλά πράγματα για το τι θα σας πω σήμερα και για τα προβλήματα των γυναικών. Η βασική ε, πρόκληση είναι η έλλειψη ενοποιημένων δεδομένων και ελπίζω πως στο μέλλον θα υπάρξει περισσότερη έρευνα για την κατάσταση των γυναικών, ειδικά των Ρωμά. Και Επίσης ε, το τι γίνεται ειδικά με τις γυναίκες. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα αναλυμένα αναγυναί με βάση το φύλλο και την εθνότητα και το εμπόδιο λοιπόν. Σύμφωνα με τα περιορισμένα δεδομένα που έχουμε φαίνεται πως οι γυναίκες Ρωμά είναι αυτές που υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις στην Ευρώπη και η κατάσταση αυτή μεγενθύνεται βεβαίω από το ότι είναι και Ρωμά και οι γυναίκες. Όπως και οι άντρε Ρωμά επηρεάζονται από την έλλειψη ίσων ευκαιριών ε, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, αποκλείονται από τι κοινωνικές υπηρεσίε και την ασφάλιση υγείας ειδικά, καθώς είναι, έχουν μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις υγείας και βέβαια αυτό ενισχύεται και από τις κοινωνικές δομές που αφορούν το φύλλο και στην ευρύτερη κοινωνία και εντός των κοινοτήτων των δικών τους. Όσον αφορά τώρα για την πρόσβαση στην υγεία, η κατάστασή τους ε, στα κράτη-μέλη τη Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι πάρα πολύ άσχημη, καθώς πάρα πολύ σπάνια κάνουν check-up και αυτό μόνο εάν αρρωστήσουν σοβαρά. γυναίκες Ρωμά με παιδιά βλέπουν τους γιατρούς πιο συχνά, αλλά αυτό μάλλον γίνεται λόγω της σκέψεων που κάνουν για τα παιδιά τους. Υπάρχει λοιπόν ένας συνδυασμός διακριτικής ε, μεταχείρισης, είναι μετά και το υψηλό κόστος νοσηλείας, οι περιπλοκές διαδικασίες και η έλλειψη εγγράφων ταυτότητας, ε, οπότε δεν υπάρχει παροχή υγείας ε, στις γυναίκες αυτές. Κατά κανόνα π.χ. στην Βουλγαρία, σύμφωνα με την έκθεση του Open Society Institute του 2008, μας δείχνει πως οι άνθρωποι με ψηλότερο κοινωνικό-οικονομικό στάτους και εκπαίδευση έχουν ε, μια καλύτερη κουλτούρα υγείας. Γύρω στο 1 τρίτο των ε, ενηλίκων γυναικών δεν έχουν ασφάλιση υγείας. 7,8 των γυναικών αυτών δεν είχαν ποτέ ασφάλιση υγείας. Στη ΔΕ Ρουμανία η έκθεση του ίδιου Ινστιτούτου την οποία ξεκίνησα εγώ όταν δούλευα στο Open Society Institute, βλέπει πως οι γυναίκες των Ρωμά αξιολογούν την δική τους ε, κατάσταση ως πενιχρή και θα λέγαμε πως 47% των γυναικών Ρωμά ε, δηλώνουν πως ε, αισθάνονται είτε άσχημα είτε πάρα πολύ άσχημα. Επίσης υπάρχει διάκριση καθώς πηγαίνουν σε ειδικές σε ειδικού θαλάμους του νοσοκομείου, τους λεγόμενους τσιγκάνικους ε, θαλάμους και στους οποίους αντιστοιχούν λιγότεροι γιατροί. Κατά τη διάρκεια λοιπόν μια συνέντευξη του Οκτώβριο 2005 ένας γιατρός ο οποίος είχε εφημερία στο μευτήριο Μισκόλτς είπε πως υπάρχουν ξεχωριστά δωμάτια πράγματι για τις γυναίκες Ρωμά αλλά αυτό ήταν για λόγους ε, υγιεινής γιατί ήταν όλες καπνίστριες. Σύμφωνα λοιπόν ε, με την έρευνα του 2005 βλέπουμε πως οι υπηρεσίε ανάγκης είναι αυτές τις οποίες χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο οι Ρωμά. Πάρα πολλοί από αυτούς αποτρέπονται και δεν χρησιμοποιούν την προληπτική ιατρική, την πρωτοβάθμια ιατρική και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Επίσης ε, δίνεται μεγάλη προσοχή στην κατάσταση όσον αφορά κάποιες χαρακτηριστικές θα λέγαμε ασθένειες των ε, Ρωμά. Το ίδιο γίνεται και σε άλλους ε, τομείς, καθώς ε, οι πολιτικές αυτές είναι εκτός του κυρίου πλαισίου της κυβερνητικής πολιτικής. Οπότε όλες αυτές οι καμπάνιες δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα όσον αφορά την ίση πρόσβαση τη υπηρεσία υγείας, γιατί δεν αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη, ειδικά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Σε κάποιες χώρες οι γυναίκες Ρωμά εξακολουθούν να ε, αντιμετωπίζουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, όπως παραδείγματο χάρη καταναγκαστικές στηρώσει ε, υφίστανται σε μεγαλύτερο ποσοστό σώματεμπορία, βία στο σπίτι και υπάρχει και γάμος ο οποίος γίνεται πάρα πολύ νωρίς και κάποιοι άλλοι παράγοντες που αποβαρύνουν την υγεία τους. Επίσης γεγονός είναι πως οι γυναίκες Ρωμά υπερεκπροσωπούνται στα θύματα της ε, σωματεμπορίας καθώς υπολογίζεται πως είναι το 80% των θυμάτων στη Βουλγαρία, ενώ στην Ουγγαρία είναι μεταξύ 40 και 80%. Όμως έχουν γίνει λίγα πράγματα για να σχεδιαστούν προγράμματα ειδικά που να αφορούν τους Ρωμά. Και ακόμα και οι γενικές πρωτοβουλίες καταπολέμησης της σώματεμπορίας δεν έχουν ε, φτάσει στους Ρωμά. Επίσης οι γυναίκες στη Σλοβακία και την Τσεχία ήταν αντικείμενο αναγκαστικής στήρωσης παρά το ότι λοιπόν αυτό σταμάτησε το 1989 εξακολουθούμε να έχουμε περιπτώσεις ε, από το, μέχρι και το 2007, από όταν μάλλον δεν έχει εξαλειφθεί η τεχνική. Το 2009 η κυβέρνηση της ε, Τσεχίας εξέφρασε τη θλίψη της στα θύματα και η Ουγγρική κυβέρνηση ε, έδωσε αποζημίωση σε ένα θύμα, όμως η Σλοβακική κυβέρνηση δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα και δεν έχει υπάρξει ένα συνολικό σχέδιο αποζημίωση των θυμάτων. Πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμιστεί ο νόμος της Ουγγαρίας για να υπάρξει μια συνένεση για στήρωση. Στη δε Ουγγαρία από 84 γυναίκες με τις οποίες κάναμε συνεντεύξεις, ο 42% δήλωσε πως ήταν θύματα βίας στο σπίτι. Η γνώση είναι όμως πως η κρατική αντίδραση είναι ανεπαρκής και ίσως να υπάρχει εδώ πέρα κάποια προκατάληψη. Παραδείγματο χάρη έρευνα Σερβία και την Ουγγαρία δείχνει πω οι γυναίκε δεν αναζητούν ιατρική βοήθεια και δεν αναφέρουν τα περιστατικά. Στην Ουγγαρία από 35 γυναίκε που έζησαν βία στο σπίτι μόνο 6 ζήτησαν τη βοήθεια τη αστυνομία. Σε μία μόνο περίπτωση θεώρησε το θύμα πώς η αστυνομία παρενεύει αποτελεσματικά. Όσον αφορά τώρα το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάποια από τα εμπόδια είναι εσωτερικά, άλλα είναι εξωτερικά. Τα πρόσφατα δεδομένα τη εκεί κυβέρνηση δείχνουν πω οι γυναίκε αυτέ είναι πιο ευάλωτε όσον και τη πιθανότητα καταλήξη σε εγκαταστάσει που αφορούν παιδιά με πνευματική υστέρηση. Η δε έκθεσή μα ε, του 2006 για τη Ρουμανία δείχνει πω υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δύο φίλων όσον αφορά την επίσημη εκπαίδευση μεταξύ γυναικών και ανδρών Ρωμά. Το δε χάσμα αυτό είναι πιο σημαντικό μεταξύ γυναικών Ρωμά και γυναικών γενικώ. 23% είναι το ποσοστό των γυναικών Ρωμά που δεν έχουν λάβει κανόση τους επίσημη εκπαίδευση. Έξι φορές ψηλότερο από αυτό που είναι στο γενικό πληθυσμό που είναι 4%. Σλοβακία, απασχόληση. Έκθεση 2007 του ΟΗΕ. έχουν περισσότερη μακροπρόθεσμη ανεργία καθώς ε, το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,6% δηλαδή συγχωρείτε απασχόληση κάτω από 5% δηλαδή επισήμως ε, δούλευαν κάτω από 5% των γυναικών παραγωγικής ηλικίας κάτω από 6% των γυναικών Ρωμά παραγωγικής ηλικία δούλευαν εκτός του νοικοκυριού. Τώρα, για την στέγαση. Η ίδια έκθεση, άμα λείπε, μας δείχνει πως ε, τα μισά αυτά, τα, μόνο τα μισά νοικοκυριά ζουν σε λιθόχτιστα σπίτια με οροφή. Μόνο οι μισοί έχουν μπάνιο, με μικρό ποσοστό επίσης έχουν τουαλέτα εντός του σπιτιού. 82,6% των ε, σπιτιών έχουν ε, τρεχούμενο νερό και 93,9% ηλεκτρισμό. Ε, σχεδόν όλα έχουν τηλεόραση, τα μισά όμως έχουν μόνο πλυντήριο. Για την δε Ρουμανία, υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων είδαν πως δεν ήταν επίσης και ε, επαρκής η αποζημίωση σε περίπτωση απαλωτρίωσης, κάτι το οποίο ιδιαίτερα τις γυναίκες. Συμπερασματικά λοιπόν οι προκλήσεις των γυναικών Ρωμα διαφέρουν από τις προκλήσεις των ανδρών Ρωμα. Οι γυναίκε και τα παιδιά λοιπόν επηρεάζονται δυσανάλογα από τη φτώχεια που επηρεάζει όλους τους Ρωμά. Το κενό μεταξύ ε, των γυναικών Ρωμά και της πλειοψηφίας των γυναικών είναι πάρα πολύ μεγάλο όσον αφορά την απασχόληση, την εκπαίδευση, την αγοραγωγική υγεία και τη γενικότερη ευημερία. Είναι λοιπόν με βάση αυτές τις ανισότητες ε, προξενεί εντύπωση το ότι δεν είχαμε περισσότερες ε, πρωτοβουλίε για να βελτιωθεί η μοίρα αυτών των γυναικών, είτε στο επίπεδο τη Ένωση, είτε στο εθνικό επίπεδο αντιθέτω. αναφέρεται αυτή η δέσμευση σε διάφορες πολιτικές και στρατηγικές όπως η στρατηγική της Λισαβόνας, η δεκαετία συμπερίληψη των Ρωμά και η πλατφόρμα του Πεκίνου. Στο εθνικό επίπεδο υπάρχουν εθνικά σχέδια καταπολέμησης των διακρίσεων, βελτίωση κατάστασης των Ρωμά, το σχέδιο αυτό της δεκαετίας και τα εθνικά σχέδια ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όμως, επειδή αυτές οι στρατηγικές δεν κάνουν συγκεκριμένη διάκριση για τις γυναίκες Ρωμά, δεν καταφέρουν να εκμεταλλευτούν το δυναμικό που παρουσιάζουν για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Μεταξύ κάποιων άλλων συστάσεων θα λέγαμε πως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να τηρήσουν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις για να μπορούν να ασκήσουν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα γυναίκες Ρωμά. Οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα όσον αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών αυτών με το να καταδικάζουν τους δράστες και όχι τα θύματα. Επίσης να αναγνωρίσουν την πολλαπλή διάκριση και να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρωμά. Επίσης όλοι οι υπάρχοντες νόμοι και οι πολιτικοί και οι μελλοντικοί νόμοι βεβαίω, να λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των φύλων και να περιλαμβάνουν διατάξεις για την αντιμετώπιση των πολλαπλών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκε που ανήκουν σε μειονότητε. Η κυβέρνηση, οι κυβερνήσει επίση πρέπει να λάβουν μέτρα για να βελτιωθεί η εφαρμογή της νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να προσπαθήσουν να τερματίσουν όλες τις διακρίσει και στον τομέα της στέγασης και της εκπαίδευση. και θα πρέπει να οργανώσουν ακροάσεις στο εθνικό επίπεδο, στα εθνικά κοινοβούλια για την κατάσταση των γυναικών Ρωμά και χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι έχουμε ακρόαση σήμερα εδώ πέρα για την κατάσταση των γυναικών Ρωμά. Για να δοθεί προτεραιότητα στις γυναίκες Ρωμά στην εθνική ε, ατζέντα και να αλλάξει ο τόνος της συζήτησης μεταξύ των πολιτικών του Γενικότερου Κοινού και του Κορσόπου Η κυβέρνηση θα πρέπει να ενθαρρύνει την οικονομική ισχυροποίηση αυτών των γυναικών θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επίστοση και να μην υπάρχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους στο σύστημα υγείας και όσες ε, γυναίκες θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, τις υπηρεσίες υγείας ε, και οι συγγενείς τους να έχουν πρόσβαση σε νομική βοήθεια. Σε στενή συνεργασία με τις ε, μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις αυτά και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν ε, σε μορφή κατανοητή προς, από το κοινό, δεδομένα αναλυμένα αναφύλλο και κοινωνική ομάδα. Και θα τελείωνα λέγοντας να διασφαλιστεί η συμμετοχή των γυναικών Ρωμά στην διαδικασία λήψη αποφάσεων. Merci, euh, Ευχαριστώ <coughs> κυρία Μιχαλασιέ για αυτή την ε, παρουσίαση σχετικά με το όραμά σας και με τις μελέτες που έγιναν σε διάφορες χώρες σχετικά με τις ε, γυναίκες ε, ΡΟΜ, πράγμα το οποίο τοποθετεί ορισμένα θέματα. Τώρα θα δώσω τον λόγο εις τις συναδέλφους μας ευρωβουλευτίνες και θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκη για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Γιανακουδάκη να μας παρουσιάσετε την, ε, ε, το θέμα σας και να κάνετε τις ερωτήσεις που θέλετε εις ε, τους στις ομιλήτριες. Ευχαριστώ. Καταρχήν δεν μ' αρέσει η ε, έκφραση ε, μειονότητα. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είμαι όμως Βρετανία, άρα μπορείτε να θεωρήσετε ότι είμαι και εγώ μειονότης. Οπότε μέσα στην ε, κοινωνία δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας ορισμός για την εθνική μειονότητα Οπότε νομίζω ότι είμαστε ευγένει υπάρξεις όπως όλοι οι υπόλοιποι. Και ε, η εθνική μειονότη σημαίνει ότι είναι μέρος ε, της ε, κοινωνίας είτε πρόκειται για άνδρες είτε για γυναίκες και όταν μιλάμε για εθνικές μειονότητες εφόσον το αναφέρετε ε, πρέπει να ε, ε, εξετάζουμε τις σχέσεις των ε, υποδεχομένων και ε, των ε, υποδεχόντων. Πρέπει να υπάρχει και από τις δύο πλευρές κατανόηση και σεβασμός. Μιλάτε για τις γυναίκες Ρομ. Είναι ενδιαφέρον γιατί δεν ήμουν καλά ενημερωμένη και νόμιζα νομίζω ότι στην Αγγλία ονομάζονται travelers, ταξιδιώτες. Εσείς μιλάτε για Ρομ Ρωμάνοι, πρόκειται μια, ε, ε, για μια εθνότητα συγκεκριμένη, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο μιλάμε για travelers και οι travelers, οι ταξιδιώτες αυτές είναι ελεύθεροι ε, και πολύ ευτυχείς ε, για την οτροπία την οποία έχουν. Έχουν βέβαια προβλήματα υγείας και άλλα διότι ε, η κοινωνία δεν δέχεται όλα τα πρότυπά τους αλλά νομίζω ότι έχουν συγκεκριμένους συνήθειες και πρέπει να τις σεβόμαστε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία κατανόηση για το που, από πού προέρχεται η κοινωνία. Πρέπει να αναφερθούμε και στις ανάγκες, αλλά ίσως αυτά είναι διαφορετικά προβλήματα από αυτά των ατόμων που είναι πιο παραδοσιακά. Θυμάμαι ότι η γιαγιά μου ε, είχε ίσως καλύτερα βότανα από οποιοδήποτε μπορούσε κανείς να βρει ε, σε φαρμακείο και υπάρχει μία ε, ε, ευάλωτη υφή την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να μπορούν να ενταχθούν, να, λάβουν, ε, να συμπεριλάβουν και τον πολιτισμό <laughs> τους, να γνωρίζει κανείς ότι πρόκειται για μοναδικές ομάδες τις οποίες πρέπει να αναγνωρίζουμε και να στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιανακουδάκη και δίνω τώρα το λόγο ε, στην κυρία Κορνέλια Ένστ για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω σχετικά με τους φιλοξενούμενους στην, ε, ε, ε, στην Γερμανία. Έχουμε μειονότητες οι οποίες ζουν εδώ και 400 χρόνια στη Γερμανία και είναι ισότιμα και ορισμένοι είναι μετανάστες που ήρθαν από την, πρώτη, την εποχή της πρώτης δημοκρατίας. Πρόκειται για ποσοστά σημαντικά 7-8 εκατομμύρια των ε, μεταναστών αυτών οι οποίοι ζουν στη Γερμανία ε, ε, πολλοί ήρθαν σαν γκάσταρμπάιτερ σαν εργαζόμενοι στη δεκαετία του 60 και υπάρχουν και πολλοί Ιουκοσλάβοι οι οποίοι τη δεκαετία του 70 ήρθαν τους υποδεχθήκαμε τότε σαν γκάσταρμπάιτερ ήρθε και η τηλεόραση για τους τους πρώτους που ήρθαν, μετά όμως άλλαξε η πολιτική και ελέγχθη ότι η Γερμανία δεν είναι χώρα για τους μετανάστες. Πολλοί από αυτούς τους μετανάστες από την Ιταλία, την Ιουγκοσλαβία, την Τουρκία έφεραν και τις γυναίκες τους, τις οικογένειές τους και ε, αργότερα ήρθαν από το Ιράν, από το Αφγανιστάν, από την Αφρική, από περιοχές που υπήρχε, υπήρχε κρίση και πολλοί ήρθαν όπως είπα και από την Τουρκία. Ε, ήρθαν και ορισμένοι ε, Εβραίοι οι οποίοι μπορούν να μείνουν υπό συγκεκριμένες συνθήκε στη Γερμανία. Αν μιλά όμως κανείς για μετανάστες πρέπει να έχει υπόψη του ότι τα άτομα αυτά έχουν δικαιώματα και ένα από αυτά είναι η κοινωνική ένταξη, ιδίω για τα παιδιά. Ε, ελάχιστοι πρέπει πρέπει να προσφέρεται και στις γυναίκες και στις μητέρες ε, ένταξη ενώ ε, όταν λοιπόν ε, μιλάμε για μετανάστες πρέπει να γνωρίζουμε τη διπλή ιδιότητα μετανάστριες αλλά και γυναίκες και ιδίω στην Ανατολική στην πρώην Ανατολική Γερμανία υπάρχει μεγάλη ανεργία για τις γυναίκες το 40% και εκεί οι μετανάστριες ζουν υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες, είναι δεμένες με τους άντρες τους και το σπίτι τους, δεν έχουν καλό ρόλο, αναγνωρίζεται μία κακώς εννοούμενη πολιτιστική παράδοση και υπάρχουν επικαλύψεις και υποχρεωτική γάμη στην Γερμανία ε, ερμηνεύεται πολλές φορές λανθασμένα η ιδέα του πολιτισμού και της παραδόσεως και οι γυναίκες ε, παραδείγματος χάρη ε, των Εβραίων έχουν δύο δυνατότητες ή να δεθούν με την οικογένειά τους είτε να αποσχεστούν. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα βέβαια. Οι γυναίκες ε, είναι θύματα σεξουαλικής βίας. Αυτό δεν είναι πρόβλημα εθνοτήτων αλλά των ρόλων των φίλων και της αποδοχής των γυναικών γενικώ. Ε, το να πάει όμως κανείς ε, στο εξωτερικό και να μεταφέρει αυτά τα προβλήματα είναι πολύ κακό. Πολλές γυναίκες από αυτές δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, δεν έχουν τις δυνατότητες να εξασκήσουν το επάγγελμά τους, οποίες ε, ε, χάνουν δηλαδή τις δεξιότητες τις οποίες έχουν και ε, παραμένουν απροστάτευτες. Πολλοί μετανάστες στην Γερμανία, μετανάστριες παραμένουν μόνο σαν γυναίκες και η ένταξη χρειάζεται και άλλες δυνατότητες να ξεπεράσει κανείς τους ρόλους των φίλων, να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των Γερμανίδων και των μεταναστριών, μη Γερμανίδων, ε, να υπάρχει κοινωνική ένταξη στην οποία δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στην Γερμανία, ιδίως όσον αναφορά τους μετανάστες. <coughs> Ευχαριστώ κυρία Ένστ για αυτή την παρουσίαση ε, της καταστάσεως στη Γερμανία και τώρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπό μας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κωνσταντίνο Φωτάκη. Κύριε Φωτάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είμαι σύμβουλος ε, του Γενικού Διευθυντή της ε, Διεύθυνσης Απασχόλησης για τα μεταναστευτικά θέματα. Πιο πολύ μπορώ να λειτουργήσω ως ακροατής ε, παρά ως αγορητής ε, στην σημερινή σας συζήτηση, γιατί εσείς έχετε πρακτική καθημερινή εμπειρία για αυτά τα ζητήματα. Θα έλεγα αρχικά πως ε, η σημερινή συζήτηση συνδέεται άμεσα με ένα λίγα ευρύτερο θέμα, δηλαδή η κοινωνική συνοχή στη μελλοντική κοινωνία των ευρωπαϊκών χωρών. Διότι τα περασμένα 15 χρόνια ε, διαπιστώσαμε μαζικές εισδροές μεταναστών στην Ευρώπη και θα συνεχιστούν αυτές οι τάσεις γιατί ε, για οικονομικούς και δημογραφικούς λόγους που προσελκύουν τους μετανάστες. Ε, στην Ευρώπη, στα σχολεία, μπορείτε να διαπιστώσετε βλέποντας τη σύνθεση των παιδιών ε, πώς θα διαμορφωθεί η πολυπολιτισμική σύνθεση της κοινωνίας στο μέλλον. Οπότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη νέα δημογραφική δομή Αλλιώς θα τεθεί σοβαρά το ζήτημα της ε, κοινωνικής συνοχής στο μέλλον. Είναι θέμα δικαιωμάτων. Ίσων ευκαιριών για όλους, είναι ηθικό το ζήτημα, αλλά είναι και θέμα επιβίωσης για την ίδια μας την κοινωνία στο μέλλον. Μιλάμε για εθνικές μειονότητες, ε, Ρώμε και άλλους και για τους μετανάστες. Υπάρχουν κοινέ πτυχές ε, αλλά και διαφορές. Αρκετά σημαντικές θα έλεγα ε, προς ε, η παρουσία της κυρίας Μιχαλάκη έκανε μια πλήρη επισκόπηση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η κοινότητα των ΡΟΜ, το πλέον ανησυχητικό κατά τη γνώμη μου σε αυτήν την δινή κατάσταση είναι το εξής. Όταν υπάρχει διακριτική μεταχείριση, δείχνουν οι μελέτες μας ότι δεν ενεργοποιούνται, δεν αναλαμβάνουν καμία δράση. Διότι είτε θεωρούν ότι ε, δεν είναι σκόπιμο, δεν ε, χρησιμεύει σε κάτι ή δεν ξέρουν σε ποιον να αποταθούν. Οπότε, για τις δράσεις και τις πολιτικές μας. Ε, ο στόχος δεν είναι μόνο να ενισχύσουμε τα δικαιώματά τους, αλλά να τους δώσουμε την δύναμη, τα εργαλεία ε, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Για την ίδια τη μετανάστευση θα έλεγα ότι το θέμα της ισότητας των φύλων έχει κέρια σημασία για τους μετανάστες, όχι μόνο επειδή ε, Υπάρχει το φαινόμενο αλλαγής της σύνθεσης ε, των μεταναστευτικών ροών, οικογενειοποίηση έτσι αποκαλείται η νέα τάση στις μεταναστευτικές ροές, αλλά έχει τροποποιηθεί και η νοοτροπία των μεταναστών και έχουν σημειωθεί αλλαγές και στην πλευρά της ζήτησης της οικονομίας. Δηλαδή, από ε, μια βιομηχανική παραγωγή περνούμε όλο ένα και περισσότερο προς τις ε, υπηρεσίες, οπότε υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον ε, για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Είναι πιο ευνοϊκός ο τομέας παροχής υπηρεσιών για την προαγωγή της απασχόλησης των γυναικών. Δοθέντως αυτού του πλαισίου θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της προάσπισης της ισότητας των δύο φύλων και η μετανάστευση συνιστά και ευκαιρία για τις γυναίκες, ε, διότι ενίοτε οι γυναίκες ε, μεταναστεύοντας ε, βρίσκουν μια ευκαιρία για να ξεφύγουν, θα το έθετα έτσι, από, τις πολιτισμι... από τους πολιτισμικούς περιορισμούς την ε, οικονομική κατάσταση της χώρας προέλευσής τους, γιατί συχνά έρχονται από χώρες ε, όπου υπάρχουν ε, πολεμικές σειράξεις ή από μια χώρα που πλήττεται από φτώχεια και πολλές περιπτώσεις γυναικών ταλαντούχων μεταναστεύοντας μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρον το κοινωνικό δυναμικό τους και να κατακτήσουν μια επιφανή θέση ε, στην κοινωνία υποδοχής. Δυστυχώς όμως ε, η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών ε, περιέρχεται σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από θέσει εργασία χαμηλή ποιότητα και αυτή τη στιγμή παγιδευτούν σε μια τέτοια θέση απασχόλησης έρχονται ε, αντιμέτωπες ε, με μια ε, κατάσταση κοινωνικού εκφυλισμού, θα το έλεγα έτσι. Παγιδεύονται λοιπόν σε αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Η ποικιλομορφία στις ομάδες των μεταναστριών γυναίκες ε, που προέρχονται, όπως μας είπε η κυρία Γκρέινερ, από την δημιουργία μιας οικογένειας, ενός οικογενειακού πυρήνα και ε, συχνά έχουν προβλήματα δικαιωμάτων, γιατί συχνά δεν έχουν το δικαίωμα ούτε καν να εργαστούν, και έχουν πολύ συγκεκριμένους ε, ρόλους που αποδίδονται στο φίλο τους συχνά που παρεμποδίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη. Κατόπιν έχουμε ένα εντελώς, μια εντελώς διαφορετική ομάδα, ε, τη δεύτερη γενιά την επωνομαζόμενη. Αυτές οι γυναίκες ε, ζουν μία διένεξη ανάμεσα σε αυτό που ζουν στο σχολείο τους, ε, στην καθημερινή τους ζωή και αυτό που βιώνουν από την άλλη πλευρά στο σπίτι τους όπου κατά πάσα πιθανότητα ζουν διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν δύο διακριτές εμπειρίες για αυτή την ομάδα γυναικών. Κατόπιν έχουμε τις τούσες άσυλο, άλλη ομάδα γυναικών, τα θύματα πολέμου, ε, γυναίκες ε, μονογονικών οικογενειών που έρχονται αντιμέτωπες με άλλου είδους ζητήματα. Θα πρόσθετα δε πως ε, σε αυτό το πλαίσιο ε, δεν βοήθησε η πρόσφατη οικονομική κρίση βέβαια, ε, διότι δεν αυξούμενη η ανεργία και αν κάνουμε ένα παραλληλισμό ανάμεσα στα ποσοστά ανεργίας ε, στις συμμεδαπές και στις μετανάστρες δηλαδή βλέπουμε ένα χάσμα 18 ποσοστιών μονάδων ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι ιδιαίτερα δε σημαντικό για τις νεοαφιχθήσεις αυτό το ποσοστό. Είναι σημαντικό να δούμε τι ισχύει για τις μετανάστες, κάνοντας τη διάκριση με ε, άλλες ομάδες ε, που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες. Ε, λοιπόν, είναι σημαντικό να δούμε ότι διαφέρει πάρα πολύ η κατάσταση ανάλογα με το αν μόλις κατέφθασαν σε ευρωπαϊκές χώρες αυτές οι γυναίκες ή αν ήδη έχουν περάσει τρία χρόνια τουλάχιστον σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι το θέμα της υποδοχής που λέγαμε των μεταναστευτικών ροών και εννοώ ότι πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες διότι Ε, η έλευση, η έγκαιρη έλευση αυτών των γυναικών έχει μεγάλη σημασία για την αξιοποίηση του δυναμικού τους. Αν δηλαδή έχουν παγιδευτεί σε χαμηλόμισες θέσεις εργασίας αυτές οι γυναίκες ενώ έχουν υψηλότερα προσόντα, ε, τότε δεν μπορούν εύκολα να διαφύγουν από αυτήν την κατάσταση. Ε, εν είδη συμπεράσματος θα έλεγα πως, ε, όπως έλεγα και νωρίτερα, πως ε, η πρόκληση είναι οι μετανάστριες και οι γυναίκες εθνοτικών μειονοτικών ομάδων ναι μεν αποκτήσουν δικαιώματα, αλλά ε, να αποκτήσουν και τα μέσα για να δραστηριοποιηθούν ρόλος που διαδραματίζουν ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ε, μόνο έτσι θα διευκολύνουμε την πρόσβαση των μεταναστών σε οργανώσεις που προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Φωτάκη για αυτή τη σύνοψη της ε, θεώρησής σας ε, για αυτό το ζήτημα, της θεώρησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το ζήτημα. Ε, εξετάσατε ολιστικά το ζήτημα, με, δηλαδή συνδέοντάς το με τον Ευρωπαϊκό Στόχο Πολιτικής Συνοχής, ε, όλοι προσπογράφουμε φυσικά αυτό το στόχο, και μας δώσατε, κάνατε και μία ιστορική αναδρομή για τις μεταναστευτικές ροές, επισημένοντα τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες ομάδες μεταναστριών. Έχουμε πρόβλημα κοινωνικό κοινωνική συνοχή ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σεβασμός ε, των ε, ε, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της χώρας προέλευσης, μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις ιστορικές περιόδους. Είπατε σήμερα βιώνουμε την οικονομική κρίση η οποία οδηγεί σε μια αυξανόμενη τάση που υφίστανται όλος ιδιαίτερος οι μετανάστριες, αλλά και γενικότερα οι μετανάστες, και το θέμα της ε, ε, Ένταση που υπάρχει διότι υφίσταται αυτή η διαφορά ανάμεσα σε όσα βιώνει μια μεταν, ε, μετανάστρια στο σχολείο και αυτό που βιώνει ενίκο. Αυτή η πολιτιστική ε, χωάνη οδηγεί ε, σε υψηλότερες ε, πιέσεις λόγω διακριτικής ε, μεταχείρισης, λόγω διαφοράς ε, των ε, βιωμάτων. Θα δώσω το λόγο τώρα στα μέλη της Επιτροπής μας που ενδεχομένως επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήσεις στα μέλη του πρώτου πάνελ. Αρχίζει η συζήτηση λοιπόν. Ποιος θα ήθελε να υποβάλει ερωτήσεις προς τους εμπειρογνώμονες. you have a uh, after that. Alors, moi, je voudrais euh, d'abord peut-être... Euh, Θα ήθελα να αρχίσω εγώ λοιπόν για να σας δώσω λίγο χρόνο ώστε να σκεφτείτε κι εσείς κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ε, υποβάλω μία ερώτηση για τις γυναίκες Ρώμα. Είχατε εμπειρίες ε, για προώθηση του αλφαβητισμού σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για τις γυναίκες Ρώμ διότι βλέπουμε ότι για να υπάρξει ένταξη πρέπει να υπάρξει αλφαβητισμός, ε, παιδεία, κατάρτιση. Τελευταία ερώτηση. Ε, που θα απευθύνω μάλλον προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και εσείς επιτόπου θα έχετε σίγουρα βιώματα, ε, ε, θέλω να θέσω το ζήτημα των επαγγελματικών προσόντων των γυναικών. Έχουμε στο μυαλό μας την εικόνα των μεταναστριών που δεν έχουν προσόντα, αλλά μιλήσατε για την παγίδα της ε, αποπροσοντοποίησης, ε, αν ε, μου επιτρέπετε τον όρο, δηλαδή όταν παγιδεύονται σε θέσεις απασχόλησης που απαιτούν χαμηλά προσόντα, γυναίκες που όμως έχουν υψηλότερα προσόντα. Ε, ποια είναι η οδός διαφυγής για αυτές τις γυναίκες και παρακαλώ να συνδέσετε αυτό το θέμα με την παιδεία και την κατάρτιση. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Η κυρία Μπάουερ τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ εις ε, την ε, ε, εκπαίδευση επίσης και αναφέρομαι στην εμπειρογνώμονα για τους ΡΟΜ σχετικά με την επιμόρφωση και την παιδεία. Στην Ανατολική Ευρώπη το βασικό πρόβλημα είναι η χαμηλή εκπαίδευση του πληθυσμού ΡΟΜ και θεωρώ ότι αυτό ισχύει για τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ίσως όχι τόσο για την Ουγγαρία. Από τη δικιά μου Πήρα όμως αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, υποκινήσει κανείς τα παιδιά των Ρώμ να μελετήσουν και να εκπαιδευτούν. Γυρίζουν στο, ε, φυσικό τους περιβάλλον και στο σπίτι δεν τους υποκινούν. Ε, η ΠΥΡΑ λοιπόν μας έχει διδάξει ότι αυτά τα άτομα Ρώμ τα οποία είναι εκπαιδευμένα δεν γίνονται αποδεκτά πλέον στην δικιά τους κοινωνία, από τους ε, δικούς τους και γι' αυτό δεν το διακινδυνεύουν. Ε, είχαμε δημιουργήσει ειδικά σχολεία ε, για εσόκλειστα παιδιά ΡΟΜ αλλά και για αυτό το πρόγραμμα και σε αυτό το πρόγραμμα οι ΡΟΜ αντιτίθενται. Ποια είναι λοιπόν η στρατηγική που θα μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε από αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ η κυρία Τόμσον. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τους ε, δύο, τις δύο μιλήτριες για την παρουσίασή τους και για τον τρόπο με τον οποίο διαχωρίζουν τις εθνικές μειονότητες από τα, τους μετανάστες οι οποίοι είναι φρεσκοφερμένοι. Ε, διότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Συνήθως οι μετανάστες εντάσσονται εις ε, τη δεύτερη τρίτη γενιά. Η γιαγιά μου ήταν Πολωνέζα και δεν είχαν τόσο ενταχθεί οι γονεί μου όσο και εγώ. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή σε πολλούς πληθυσμούς και πολλές φορές το πρόβλημα των Ρώμη είναι ότι πρέπει να τους αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις και ε, ένα μεγάλο ποσοστό ρομ. Εάν όμως μελετήσετε την Ευρώπη θα δείτε πόσο πληθυσμοί έχουν ενταχθεί. Στη Δανία δεν είχαμε ποτέ ε, ρομ ελάχιστους μόνο, ε, διότι ε, πριν από δύο αιώνες οι Ρώμ εστάλθηκαν στην Σουηδία και στη Σουηδία εντάχθηκαν, αλλά στην δεκαετία του 60 η κυβέρνηση της Σουηδίας προσπάθησε να εντάξει τους Ρομ που τώρα έχουν ενταχθεί, αλλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το συζητήσουμε ε, αν είναι ε, μία ε, ένταξη ή ε, μία αφομοίωση, δηλαδή αν έχουν διατηρήσει τις παραδόσεις τους, ποια είναι η στρατηγική για να μπορέσουν οι Ρώμ να ενταχθούν. Και στην Ισπανία έχουμε δει ότι έχουν ενταχθεί πολύ καλά. Άρα όλα εξαρτώνται από τα μέτρα που λαμβάνονται. Είμαι όμως πολύ ευτυχής ότι ε, ο Επίτροπος για Απασχόληση και Κοινωνική ε, Ενσωμάτωση έχει ζητήσει να καταρτιστεί μία ομάδα και ελπίζω ότι θα έχουμε και στατιστικές για να μελετήσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τόμσον. Αν δεν υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να λάβει το λόγο, σας προτείνω να δώσουμε το λόγο ή στην εισηγήτρια. Η πρώτα στην κυρία συγκυρια κυρια μιελαχε για όλα αυτά τα προβλήματα των ΡΟΜ που βλέπουμε ότι είναι στο επίκεντρο των ε, ε, της συλλογιστικής μας. Δεν πρέπει να αναφερθούμε μόνο εις την κοινότητα των Ρώμα, αλλά να έχουμε μια σφαιρική αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ καλές οι ερωτήσεις. Θα τις πάρουμε τη σειρά. Θα αρχίσω με τα δικά σας σχόλια, διότι Μιλήσατε για την διαφορά ανάμεσα στους Ρώμε και τους τράβελες, τους οδηπόρους, τους ταξιδιώτες. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες όντως. Έχουμε τους τράβελες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Έχουμε τους Αθήκανους στο Κωσυφοπαίδιο, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια εθνοτική ομάδα, αλλά αυτό αποκαλούνται έτσι. Και εξαρτάται αν ανήκουν σε παραδοσιακέ κοινωνίε ή σε κάποιο αστικό περιβάλλον. Αληθεύει αυτό. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, θα έλεγα, ή και για τι υπόλοιπε χώρε όπου διαμένουν, έχουν προβλήματα όπως αναφέρατε. Πέρσι τον Οκτώβριο δημοσιεύτηκε μία μελέτη ε, για το πρόβλημα στέγασης που έχουν, ε, παραδείγματος χάρη, και επιτρέψτε μου να διαβάσω τι λέει η μελέτη. Πολλοί τράβελες που ε, διαμένουν παράνομα σε καταβλισμούς χωρίς καμία πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και δεν είναι ιδιοκτήτες ε, και έχουν κατασκευαστεί καταβλισμοί χωρίς ε, καμία άδεια πολεοδομίας ε, και αυτό οφείλεται σε έλλειψη οποιασδήποτε άλλη στέγαση. Να λοιπόν ένα πρόβλημα που έχουν. Δεν έχουν άδεια διαμονής και πρέπει να μετακινούνται διαρκώς και αυτό φυσικά σχετίζεται με το πρόβλημα παιδείας για τα παιδιά τους και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Για τις λοιπές διαφορές που αναφέρατε ανάμεσα στους δρόμ και τους μετανάστες, ε, ε, το θέμα των δρόμων υπάρχει εδώ και αιώνες. Και όταν αναφερόμαστε στους δρόμ ε, με τον όρο μειονότητα, είναι λίγο πλημελές γιατί θα μπορούσαν να συνιστούν και ε, πλειοψηφία, εάν ε, συνενωθούν όλοι οι ρόμ που υπάρχουν σκορπισμένοι στην Ευρώπη. Ειδικά όταν μιλάμε για κάποιες βαλκανικές χώρες. Μιλάμε φυσικά για τις ίσες ευκαιρίες, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η πρόσβαση ε, στα βασικά δικαιώματα που αρνούμαστε στους ΡΟΜ. Επανερχόμεθα λοιπόν στο κέριο θέμα. Είναι απαράδεκτο να ε, συζητούμε για κάποιους που δεν έχουν ταυτότητα και άρα δεν έχουν και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, ε, δεν μπορούν να διεκδικήσουν βασικά δικαιώματα. Και γι' αυτό επανέρχομαι στα θέματα των δεδομένων. Έκανα αυτή την παρουσίαση γιατί αντικατέστησα μία συνάδελφό μου και αποφάσισα να μιλήσω για τα δεδομένα. Ευτυχώς έχω και εγώ συγκεκρι... κάποιες εμπειρίες ε, στον τομέα αυτό. Και παρόλα τα δεδομένα που έχουμε, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση επιτόπου και δύσκολα μπορούμε να υποθέσουμε ε, τι βιώνουν οι γυναίκες σε Οπότε το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να συλλέξουμε δεδομένα για να γνωρίζουμε ακριβώ πώ έχει η κατάσταση. Για τα προγράμματα τώρα αλφαβητισμού, εμεί στο κέντρο μα δεν έχουμε τέτοια προγράμματα. Γιατί ο στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των γυναικών και να προωθήσουμε την πρόσβασή τους στις βασικές υπηρεσίες. Ε, τα προγράμματα αλφαβητισμού είναι ε, δουλειά μη κυβερνητικών οργανώσεων, ειδικών οργανώσεων, που διαθέτουν και τα απαιτούμενα μέσα για να προστατεύεται η γλώσσα των Ρώμε. Για ε, τα χαμηλά προσόντα τώρα, το άλλο θέμα που έθιξε η κυρία Μπάουερ, φυσικά είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο. Αληθεύει αυτό. Και είναι πολύ πολύμορφες ε, οι προκλήσεις. Ε, γιατί δεν περιορίζονται μόνο στο σχολείο, αλλά υπάρχουν και στην κοινωνία. Ε, διακριτική μεταχείριση στην εκπαίδευση, παραδείγματο χάρη. Αν δεν υπάρχει το πρωτογενέ δικαίωμα πρόσβαση ε, στην παιδεία, οποιαδήποτε παιδεία, οποιοδήποτε επίπεδου, ε, η διακριτική μεταχείριση δεν έχει καμία σημασία γιατί ναι, πρόκειται για δασκάλους ε, που δεν έχουν τα πετούμενα προσόντα, δεν πηγαίνουν τα παιδιά στα μαθήματα, είναι σε ε, ε, κρανίου τόπος, στείνονται αυτοσχέδια κάποια μαθήματα που δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Και διαπιστώνουμε λοιπόν διακριτική μεταχείριση. Στην Τσεχία, παραδείγματο χάρη, τεκμηριώνεται αυτό το πρόβλημα γιατί ε, δείτε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, όπου αναφέρεται το πρόβλημα που υπάρχει στην ε, Τσεχία και θεωρούνται τα παιδιά Ρομ ως καθυστερημένα. Στη Ρουμανία επίσης υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα σοβαρά προβλήματα διακριτικής μεταχείρισης ε, στην παιδεία. Οπότε ε, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να ε, προσφέρουμε ποιοτική πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και αυτό μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Βουλγαρία και εδώ έχουμε εκπρόσωπο της Βουλγαρίας εδώ και 7 χρόνια οι ΜΚΟ μικρών ε, εργάζονται για να ασχοληθούν Παραδείγματο χάρη με τα λεωφορεία που θα πηγαίνουν τα παιδιά κάθε μέρα στο σχολείο και πάνε τα παιδιά, σηκώνονται το πρωί, πηγαίνουν ε, στο σχολείο. Αλλά παρόλη αυτή την προσπάθεια δεν είχε στενιστεί αυτή την πρακτική η κυβέρνηση για να τη μετατρέψει δηλαδή σε κυβερνητική πολιτική και ε, παρέχουμε κάποια λεωφορεία αλλά όχι για όλα τα παιδιά που το χρειάζονται. Υπάρχει δηλαδή η βούληση των γονέων και των παιδιών, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να συνεργάζεται και η κυβέρνηση. Ε, είναι, πρέπει να υπάρχει διμερής προσέγγιση από την κυβέρνηση και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, για τις μετανάστριες τώρα, για τους μετανάστες μάλλον και τις διαφορές που έχουν από, ε, σε σχέση με τους ΡΟΜ. Ναι, έχουν ειδικέ ανάγκες οι ΡΟΜ και σε κάποιες χώρες ε, από υπήρξε μια προσπάθεια να ενταχθούν οι Ρώμα, αυτό που είπατε για τη Σουηδική κυβέρνηση. Ναι, ήταν ιδιαίτερα προδραστική η Σουηδική κυβέρνηση για να προστατεύσει γενικότερα τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων, ε, των γυναικών ε, και αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα η γλώσσα του στη Σουηδία και διαφυλάτεται ο πολιτισμός του στα σουηδικά σχόλια. Παρόλα αυτά, ε, εξακολουθούν να υφίστανται διακριτική μεταχείριση για την πρόσβαση σε κάποια δικαιώματα, κυρίως ως προς τη στέγαση. Ε, είναι πιο δύσκολο για ένα ρομ, παραδείγματος χάρη, ε, να να ενοικιάσει ένα διαμέρισμα, παραδείγματο χάρη, γιατί υπάρχει διάκριση από την πλειοψηφία στην ε, κοινωνία για να ε, ενοικιαστεί ένα διαμέρισμα στο ΡΟΜ. Βέβαια γίνονται κάποια βήματα και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της ε, Σουηδίας αντίστροφα. Δηλαδή όταν για την αναγκαστική στήρωση υπάρχει αποζημίωση σε χώρες όπως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, τότε ε, θα πρέπει να συνεργαστούν αυτές οι κυβερνήσεις με την ε, Σουηδική κυβέρνηση και να αντιγράψουν αυτές τις καλές ε, πρακτικές. Νομίζω ότι απάντησα σε ερωτήσεις σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα θέλατε κι εσείς εντάχει παρακαλούμε να σχολιάσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Τρία λεπτά το όριο κυρία Γκράνε. σας παρακαλούμε. Uh, είπα και προηγουμένως, ε, είμαι ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταναστών και ε, εργαζόμαστε εις ε, τη βάση. Έχω εργαστεί για τις Αφρικανές γυναίκες στην Γερμανία και οι συνάδελφοί μου έχουν συνεργαστεί και με άλλες ομάδες και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη, υπάρχουν πολλές διακρίσεις εναντίον τους και οι γυναίκες αυτές δεν ε, εντάσσονται χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Ε, ντρέπονται, βρίσκονται σε ένα πλαίσιο που δεν τους ταιριάζει. Υπάρχει πρόβλημα ε, οικιστικό, υπάρχει πρόβλημα εργασίας, πρόβλημα του χρώματος του δέρματος και αυτό το βλέπετε και στη δεύτερη και την τρίτη γενιά όπου υπάρχει μία σύγκρουση. Όσο λοιπόν δεν επεμβαίνουμε και να συζητήσουμε αυτή, αυτά τα θέματα, εγώ προσπαθώ να συνεργαστώ, αλλά ο καθένας τραβάει από τη δικιά του μεριά και πρέπει να βοηθήσουμε την κοινότητα αυτή να ενταχθεί, αλλά θα πρέπει και η κοινωνία των ε, δεκτών να δεχθεί αυτή την ε, ε, την ε, ε, συνεργασία διότι τα παιδιά γεννιούνται στη Γερμανία αλλά ή ψάχνουν ποια είναι η ταυτότητά τους ή λένε πότε θα πάμε πίσω στην Αφρική δεν έχουν πάει ποτέ στην Αφρική οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα για να κάνουν αυτό το ταξίδι σέρνονται από το, τη μία χώρα στην άλλη και ε, όταν φύγαμε από τη χώρα μας είχαμε έναν πολιτισμό, είχαμε παραδόσεις και εάν δεν ε, συνεργαστεί η κοινωνία τότε οι μετανάστες όταν μετακινούνται σε μια άλλη χώρα κρατούν τις, τις αρχές τους και τις παραδόσεις τους όπως η γεννητικοί ακροτηριασμοί ή τη θέση της γυναίκας και του άντρα και ε, εάν δεν μπορέσουν να ενταχθούν τελικά γυρίζουν στη χώρα από την οποία προήλθαν. Νομίζω ότι ε, δεν μου δώσετε περισσότερο χρόνο, εγώ θα είχα πολλά ακόμη να σας πω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φωτάκης. Νομίζω πως ε, πρέπει να απαντήσω σε αυτό το ερώτημά σας για τα προσόντα και αυτό το οποίο εμείς λέμε σπατάλι εγκεφάλων. Μας ρωτήσατε ποιοι τομείς ε, επηρεάζονται από αυτό το φαινόμενο. Προφανώς θα έλεγα η υγεία στα νοσοκομεία μας Έχουμε πολλούς γιατρούς από τρίτες χώρες, αλλά και από χώρες από την, όπως η Πολωνία, που, που δουλεύουν, με συγχωρείτε, ως νοσηλευτές. Και την, την νυχτερινή βάρδια κιόλα. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν. Το πρώτο θέμα είναι η αναγνώριση των προσόντων και αυτό είναι πραγματικό ζήτημα. πώς θα υπάρξει ισοδυναμία μεταξύ ενός πτυχίου από τη Μογγολία ή το Βιετνάμ. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Και δεν ξέρετε πως ε, για να υπάρξει ισοδυναμία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε μεγάλες δυσκολίες και αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της Κομισιόν προσπαθούμε και η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Εκπαίδευσης και Απασχόλησης και νομίζω πως θα έχουμε πρόοδο τα επόμενα χρόνια ουσιαστική αλλά είναι πολύ σημαντικό ζήτημα επιπλέον Υπάρχει πέρα από τα πτυχία το ζήτημα του να μπει γνώση στο πλαίσιο της χώρας υποδοχής. Γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές. Πρώτα απ' όλα η διαφορά της γλώσσας και όταν δουλεύει κανείς ειδικά σε πολύ εξειδικευμένες δουλειές έχει μεγάλη σημασία η ακρίβεια. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί μετά το θεσμικό πλαίσιο. Όσοι δουλεύουν πρέπει να ξέρουν το θεσμικό πλαίσιο της χώρας υποδοχής που είναι ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, διαφορετικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει αρκετές δράσεις και σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας μιλάμε για 600.000 άτομα. Είτε μετανάστες είτε άνθρωποι που ανήκουν σε μειονότητες που είναι δικαιούχοι κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επίσης όταν παγιδευτούν σε τέτοιες δουλειές χαμηλών προσόντων δύσκολα φεύγουν από εκεί γιατί συχνά τους εκμεταλλεύονται εκεί πέρα τον προηγούμενο μήνα ήμουν σε ένα συνέδριο των EuroCities στο Λονδίνο και είχα μια ομάδα εργασία ακριβώς για αυτό το ζήτημα και εκεί πέρα υπήρχαν διάφορες ΜΚΟ και οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν πάρα πολλέ ώρε στι δουλειέ αυτέ και το να λείψουν έστω και μία μέρα για να πάνε συνέντευξη σημαίνει ότι θα χάσουν τι δουλειέ του. Κάτι το οποίο δεν γίνεται γιατί ε, τα έξοδα τρέχουν, οι μισθοί του είναι πολύ χαμηλή. Οπότε δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν ε, τις, ε, πιθανό, τις δυνατότητες που υπάρχουν για να βρεθούν σε μια καλύτερη δουλειά. Οπότε όλες αυτές είναι πτυχές που ενισχύουν το φαινόμενο αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Φωτάκη. Ευχαριστώ κύριε Φωτάκη. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Μπρίτα Τόμσεν, η οποία είναι η σκιώδης εισηγήτρια. Όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ για ε, την, ε, ε, τα σχόλιά σας κύριε Φωτάκη. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ομάδα συζήτησης. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις παρεμβαίνουσες και θα καλούσα τις υπεύθυνες για το δεύτερο πάνελ να έρθουν στο βήμα η κυρία Ελίζαμπεθ Μέλλερ Γένσεν, ο κύριος Κεμάλε Γιούπ για να ξεκινήσουμε το δεύτερο πάνελ σχετικά με τις πρακτικές ένταξης. Και μετά η κυρία Τόμσεν θα λάβετε το λόγο. Donc nous allons voir maintenant Λοιπόν, τώρα θα ασχοληθούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα ένταξης. si Donc λοιπόν αμέσως τον λόγο στην κυρία Μέλλερ Γένσεν του Δανικού Κέντρου Ενημέρωση σχετικά με τις γυναίκες και τη διάσταση του φύλου ε, στην Δανία και θα μας μιλήσει για τις ε, πολιτικές ένταξεις στη χώρα της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την πρόσκλησή σας με ανυπομονησία την ευκαιρία αυτή να σας μιλήσω και μόλις συνειδητοποιήσω ότι μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου. Οπότε αυτό θα κάνω. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω το δίκτυο Κβίνφο που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τις γυναίκες ε, που έχουν μεταναστεύσει, είναι πρόσφυγες ε, και συγκρίνει με τις ε, γυναίκες της γηγενής στην Δανία. και διαπίστωσα πως ε, είχαμε επιτυχία όταν ε, μια γυναίκα μας είπε πως μεντοράς μου ή μεντοράς μου είναι θα έλεγα το ανθρώπινο GPS μου και εκεί πέρα λέω πραγματικά κάνουμε τη δουλειά μας οι καθοδηγητές αυτοί που έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να κατευθύνουν αυτές τις γυναίκες αλλά πρώτα απ' όλα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες ε, για το Κουδίνφο. Το Κουδίνφο είναι ένα κέντρο πληροφόρησης ε, για την ε, ισότητα των εθνοτήτων που ξεκίνησε στην δεκαετία του 60 στη Δανία. Είναι ένα εδρεωμένο ίδρυμα που υπάγεται στο Υπουργείο πολιτισμού έχουμε λοιπόν ήδη ε, σε όλους τους τομείς της ε, κοινωνικής ζωής και τα τελευταία δέκα χρόνια προσπαθήσαμε να επεκταθούμε στο ίντερνετ, ξεκινήσαμε μια εγκυκλοπαίδεια με βιογραφίες αξιόλογων γυναικών στην ε, Δανία, τα βγάλαμε όλα αυτά στο διαδίκτυο, έχουμε επίσης την ιστορία των γυναικών της Δανίας που μπήκε και αυτή στο διαδίκτυο και ένα διαδικτυακό περιοδικό, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες ε, που αισθάνονται ότι έχουν μια σχέση με το ίδρυμα αυτό μπορεί να μας παρακολουθήσουν και μέσω Twitter οπότε το 2003 είχαμε την ιδέα που ήταν και πρόκληση για τα δίκτυα που ασχολούνται με τις γυναίκες να ενεργοποιηθούν και να δούμε πώς ε, θα χρησιμοποιήσουμε με τον καλότερο τρόπο το δίκτυο αυτό του Κβίνφο και, στην αγορά εργασίας. Ξεκινήσαμε με ένα μικρό ε, έργο με 12 μέντορες ε, δεν ήμασταν. Δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τους μετανάστες ε, στην Δανία, αλλά όταν ε, έστειλαν αυτό το email, εκατοντάδες γυναίκες θελοντικά είπαν πως θέλω εγώ να γίνω μέντορας και αμέσως είχαμε επιτυχία. Το επόμενο έτος λάβαμε δύο βραβεία. Ένα βραβείο από την, από ένα γυναικείο περιοδικό της ε, Δανίας και άλλο ένα βραβείο επίσης. Οπότε ήταν ε, mentors που ήθελαν να δώσουν συνεντεύξεις, να πούν τις εμπειρίες τους. Μιλάμε για πάνω από 5.000 γυναίκες ε, μετανάστριες που έλαβαν μέρος. Οπότε είχαμε πάνω από 2.000 ζευγάρια που ήρθαν. Είχαμε γραφεία σε τέσσερα σε τέσσερις πόλεις, ε, γυναίκες που προέρχονται από 127 χώρες, ε, γυναίκες με πάρα πολλά προσόντα που βρήκαν δουλειές γιατί ήταν τόσο ικανές, είχαν τόσα προσόντα και είναι ένα από τα λίγα έργα μας που ήταν τόσο επιτυχή όσον αφορά δηλαδή την έβρεση εργασίας γιατί βεβαίως δουλειά έβρισκαν, αλλά δεν ήταν πάντα η κατάλληλη δουλειά. Εάν έχει λοιπόν κανείς έναν μέντορα, συνήθως είναι γυναίκες που κάνουν την ίδια δουλειά, π.χ. μία γιατρός, μία νοσοκόμος, για τον αντίστοιχο άνθρωπο που συμβουλεύει και μπορεί να του πει πολύ εξειδικευμένο τι γίνεται και με τα προσόντα, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να βρουν δουλειά αυτές οι γυναίκε Γιατί και στο ε, προηγούμενο, στο γραφείο είχαμε ένα γραφείο ε, κοντά σε οικίε που ήταν τα λεγόμενα γκέτο των μεταναστών στο Βαλσιμόζε παραδείγματος χάρη κοντά στην ε, Κόπενχάγη οπότε τους είχαμε μια κοινωνική μέντορα η οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι εκπαιδευμένοι είτε σε κοινωνικές επιστήμες, οπότε δεν είχαμε μόνο κοινωνιολόγους ή ανθρωπολόγους, αλλά το βασικότερο μια γυναίκα, μια γυναίκα που ενδιαφέρονταν και συνεργάζονταν πάρα πολύ στενά μαζί τους και είχαμε και άμεσα αποτελέσματα. Οπότε Αρκετοί το κάνουν εθελοντικά, είναι αυτό το οποίο λέμε value-based, υπάρχει δηλαδή μια αλληλεγγύη, προσπαθούν οι γυναίκες να βοηθήσουν μια άλλη γυναίκα, να την ενσωματώσουν στην κοινωνία της Δανίας. Θέλουν λοιπόν να λάβουν μέρος σε κάτι το οποίο έχει τις ίδιες αξίες με αυτές και αφορά την ισότητα, το να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κοιτάξουν τους άλλους ως ίση και βλέπουμε και τι μοιραζόμαστε με γυναίκες ε, ε, που έρχονται από άλλα μέρη του κόσμου στην ε, Δανία. Αλλά βέβαια αυτή είναι και μεγάλη διαφορά το να ήταν κάποιος επαγγελματίες. Βλέπουμε πως υπάρχει αυτό το mentoring που ξεκίνησε σε μεγάλες επιχειρήσεις στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και αλλού Είχαμε και συμβάσεις τις οποίες όριζαν δηλαδή τι στόχους έχουν, τι ήθελαν να κάνουν ε, και μετά βλέπαμε ανατακτά διαστήματα το τι γίνονταν και το τι πρόοδο είχαν επιτύχει και ήταν σημαντικό αυτό ε, καθώς ενδιαφέρονταν οι γυναίκες ε, με πάρα πολλά προσόντα, επαγγελματίε κτλ. Και οι μέντορες ε, αυτοί μετά έδωσαν και μια συνέντευξη μιας ε, ώρας ε, για να μπορέσουν να βγάλουν, αν θέλετε, κάποιους κάποιες παροπίδες πολιτισμικές με τις οποίες έβλεπαν τα τα πράγματα, να μην βλέπουν ε, την εμφάνιση των ανθρώπων, το πώς είναι ντυμένοι, αλλά να δουν πραγματικά τι προσόντα έχουν αυτές οι γυναίκες, ε, γιατί ήρθαν, τι θέλουν να κάνουν στη Δανία, ποια είναι τα όνειρα, οι ελπίδες τους, τι ελπίζουν από τη ζωή στη Δανία. Και πραγματικά το αναπτύξαμε αρκετά καλά. Υπάρχουν και άλλα επίπεδα που προστέθηκαν σε αυτό, παραδείγματος χάρη ε, είχαμε την δεύτερη γενιά μεταναστών που ήταν πραγματικά πάρα πολύ ικανοί. Στην αρχή δεν υπήρχε τόσο ενδιαφέρον, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορέσουν να βοηθήσουν τους νέους μετανάστες. Ε, και να δεχτούν σε όλο αυτό το δανειζικό δίκτυο και μετά βλέπουμε το τι μπορεί να επιτύχει ένα ισχυρό δίκτυο και να αναπτύξει ένα πολιτικό πρόγραμμα, δηλαδή πιο το ότι μετά 15 ισχυρές ε, πολιτικοί, π.χ. η κυρία Μπρετατόμισεν, ε, ασχολήθηκαν ε, με αυτό το θέμα και είχαμε 15 λοιπόν νέες μετανάστριες που θέλουν να κάνουν καριέρα στην Δανία και τις φέραμε σε επαφή με τις μέντορες αυτές και παραδείγματος χάρη είχαμε την εκατοστή επέτειο του δικαιώματος ψήφου των γυναικών ε, στην ε, Δανία και εκεί πέρα με αυτή την ευκαιρία γνώρισαν πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, μετά είχαμε στο Βαλσμόζε πάλι και στο Όντζε νέους που με χρηματοδότηση ενός ιδιωτικού ταμείου πήγαν σε ένα σχολείο και βρήκαν έναν δανό μέντορα που τους ε, υποστήριζε στην εκπαίδευση γιατί αυτό είναι μια στήριξη που δεν υπάρχει στην ε, οικογένειά τους. Γιατί δεν υπήρχαν και απαραίτητες επαφές ε, στην Δανέζικη κοινωνία. Οπότε τώρα είχαν αυτή την υποστήριξη, υπήρχε και απαραίτητη χρηματοδότηση για να απτυχθεί αυτό το έργο με τους, με τους ε, δεν ξέρω αν έχω άλλο χρόνο. Θα μπορέσουμε να ε, συμπληρώσουμε και δεδομένων των ερωτήσεων που θα κάνουν οι συνάδελφοι θα υπάρξει και συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εμπειρία της Δανίας και είμαι ε, σίγουρη ότι θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, ε, ε, ερωτήσεις να σας κάνουμε. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Κεμάλ Λεγιού, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την Προστασία κατά της διάκριση τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και θα θέλαμε να ακούσουμε την εμπειρία σας. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα να κάνουμε την παρουσίασή μας για την ένταξη των γυναικών που ανήκουν σε μενοτικές εθνοτικές ομάδες. Δεν θα μιλήσω για τις μετανάστριες στη Βουλγαρία, διότι είναι αμεληταίο ε, το ποσοστό τους. Η ισότητα των δύο φίλων στη Βουλγαρία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα ε, και ε, από τον νόμο κατά της διακριτικής ε, μεταχείρισης στην αγορά εργασίας. Αλλά δεν υπάρχει νόμος που να ενθαρρύνει την συμμετοχή αυτών των γυναικών στην πολιτική και πολιτισμική ζωή. 15% των γυναικών στην Βουλγαρία Ε, είναι άγνωστες. Δεν γνωρίζουμε την ηλικία τους, ε, την, ε, τα στοιχεία ως προς την απασχόλησή τους, ε, τους κινδύνους που διατρέχουν για οικογενειακή βία. Υπάρχουν πολλές πτυχέ που δεν γνωρίζουμε διότι δεν έχουμε συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα στη διάθεσή μας και αυτό εξηγεί και την απουσία μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Η Επιτροπή Προστασίας κατά της διακριτικής μεταχείρισης έχει δεδομένα που δείχνουν πως οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονοτικές εθνοτικές ομάδες υφίστανται διαφόρων ειδών διακριτικές μεταχειρήσει ε, λόγω του φύλου και λόγω της εθνοτικής τους και σε μια περίοδο ε, οικονομικής κρίσης ε, οι γυναίκες αυτές ε, είναι και οι ευπαθέστερες, είναι οι πρώτες που χάνουν τις θέσεις απασχόλησής τους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και πολύ συχνά αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια ε, στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην κοινωνία. Προτείνουμε να ε, δρομολογήσουμε μία ε, διαδικασία ενσωμάτωσης της διάστασης της ότας των δύο φίλων σε όλες τις πολιτικές για να τις ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν σε, στα κοινωνικά δρόμενα και για να αναβαθμίσουμε τη θέση τους. στις εκλογές, ε, σε ευρωπαϊκές ε, εκλογές ε, στη Βουλγαρία και στις εθνικές εκλογές οργανώθηκε μία εκστρατεία σε συμμετοχή αντρών και γυναικών και είχαμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 40% των βουλευτών από τη Βουλγαρία είναι γυναίκες. τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή μάλλον όχι τα ίδια αλλά αντίστοιχα 20% των ε, γυναικών συμμετέχουν στην τωρινή ε, κυβέρνηση, βελτίωσε σε σχέση με, ε, τις προηγούμενες, με την προηγούμενη κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, Μόνο 1% των γυναικών εκπροσωπούν τις μειονοτικές θεντοντικές ομάδες στο κοινοβούλιο μας. Στη βουλγαρική κυβέρνηση το 17% των μελών της κυβέρνησης είναι γυναίκες και έχουμε την πρώτη πρόεδρο επίσης ε, του Εθνικού Κοινοβουλίου που είναι γυναίκα. Λόγω της απουσίας αυτής ε, των στατιστικών δεδομένων ε, για τις μειονοτικές εθνοτικές ομάδες έχουμε μια ομιχλώδη μάλλον η εικόνα της κατάστασης και δυσχεραίνονται οι προσπάθειες που καταβάλουμε για να τονώσουμε την ένταξή τους ή για να παρακολουθήσουμε τα μέτρα που έχουν ήδη αναλυθεί και κατά πόσο έχουν αποτέλεσμα. Ε, ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουμε ιδιαίτερες δυσκολίες διότι πρέπει να προστατεύονται τα ατομικά δεδομένα, αλλά είναι απαρέγκλητη ανάγκη να συλλέξουμε ε, δεδομένα, ούτω ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τι συμβαίνει με την νομική υπόσταση των γυναικών που ανήκουν σε μειονοτικέ ε, ομάδε, ε, να διαπιστώνουμε ποια είναι τα ποσοστά ανεργία σε αυτέ τι ομάδε και να χρησιμοποιήσουμε και τα δεδομένα τη Eurostat, τόσο ώστε να διαμορφώσουμε μια πληρέστερη εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο, απουσία δηλαδή στατιστικών δεδομένων, αναδύονται διάφορες ε, δυσκολίες ε, για αυτές τις ε, μειονοτικές ομάδες και δεν καταφέρνουμε να ρυθμίσουμε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πολύ συχνά οι πολιτικές που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ε, υπόστασης των γυναικών Ρώμα, παραδείγματος ε, χάρη, οφείλονται στην παραγνώριση των δικαιωμάτων από τις ίδιες τις γυναίκες ε, ΡΟΜ. Οι μειονοτικές ομάδες στην Βουλγαρία που εκπροσωπούν 15,6% του πληθυσμού που και το μεγαλύτερο κομμάτι έρχεται από την Τουρκία και το 51,6% είναι γυναίκες. Στις ε, ομάδες ε, των Τούρκων και των Ρώμ Υπάρχουν περισσότεροι άντρες ε, παρά γυναίκες ε, και δείχνουν δημοσκοπήσεις ότι οι εθνικές στρατηγικές ε, καθώς και τα προγράμματα που υλοποιούνται από, τις, από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεν λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των ομάδων, παραδείγματο χάρη στον τομέα της παιδείας. Πολύ συχνά τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες παραδόσεις αυτών των ομάδων τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Συχνά οι γονείς φοβούνται να ε, στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο σε ένα άλλο χωριό, γιατί στο δικό τους δεν υπάρχει σχολείο, παραδείγματος χάρη. Αυτό ναι, σχετίζεται φυσικά με την ύπεθρο περισσότερο παρά με το αστικό περιβάλλον. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα, κυρίως για τους Ρώμα και τους Τούρκους. Ένα τέταρτο των Ρώμων στη Βουλγαρία είναι αναλφάβητοι. Να επισημάνω δε ότι ε, στα δέκα πρώτα χρόνια μετά την πτώση του κομμουνισμού και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, αυτό το φαινόμενο του αναλφαβητισμού διωγγώθηκε ε, σε ανησυχητικά επίπεδα. Από αυτή την πλευρά λοιπόν θα έλεγα πως ε, οι γυναίκες πλήττονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άντρες λόγω το εκπαιδευτικού τους ε, επίπεδου. Ο αναλφαβητισμός αυτός ε, που εκδηλώνεται σε άγνοια των γονέων οδηγεί και σε μια έλλειψη βούλησης στα παιδιά να παρακολουθήσουν μαθήματα στο σχολείο. Χρειάζεται λοιπόν να αναλάβουμε ειδικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συγκεκριμένες περιστάσεις για να εξασφαλίσουμε τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών. Η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική αν πρόκειται αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πολύ συχνά ε, δεν μπορούν οι ΡΟΜ να απασχοληθούν και ε, προβάλλεται ως επιχείρημα το χαμηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο, τα χαμηλά τους προσόντα και τα δέκα τελευταία χρόνια η ανεργία πλήττει ολόκληρη την κοινότητα των ΡΟΜ που δεν έχουν πλέον την δυνατότητα να εγγυηθούν μια σωστή εκπαίδευση για τα παιδιά τους, να τους ε, μεταβιβάσουν μια αίσθηση ευθύνης, κοινωνικής ευθύνης και να τους δώσουν μια ουσιαστική δυνατότητα να ενταχθούν μετέπειτα στην κοινωνία στην οποία ζουν. Οι γυναίκες Ρώμα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας λόγω της οικογενειακής τους κατάστασης. Υπάρχουν προκαταλήψεις κατά των γυναικών Ρώμα, συνήθως έχουν πολλά παιδιά και πολύ συχνά δεν γνωρίζουν ποιες δυνατότητες έχουν και μπορούν να εκμεταλλευτούν στην αγορά εργασίας. Στην ε, Βουλγαρία ε, Συχνά οι γυναίκες ε, ΡΟΜ εργάζονται σε θέσεις όπου δεν απαιτούνται καθόλου προσόντα ή εργάζονται και στην μαύρη οικονομία, στην παραοικονομία. Η εγκληματικότητα είναι διαδεδομένη δυστυχώς ε, κυρίως στις πόλεις. Ε, η εθνική πολιτική τώρα του Υπουργείου Απασχόλησης ε, για να προαχθεί η θέση τους στην αγορά εργασίας δεν έχει τελεσφορήσει μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά και το κοινωνικό τίμημα που καταβάλουμε είναι ιδιαίτερα υψηλό, κυρίως για τις ε, γυναίκες δρόμου που έχουν ε, μόνογονεικές οικογένειες, ε, μονογονεϊκές οικογένειες με πολλά παιδιά που συχνά υποχρεώνονται να καταφύγουν στην πορνεία για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν για τις ίδιες και τα παιδιά τους. Αντίθετα, η τουρκική μειονότητα ζει μια διαφορετική κατάσταση, αντιμετωπίζει διαφορετικές ε, δυσκολίες. Ε, έχουν ε, καλύτερη παιδεία, αλλά υπάρχουν παρόλα αυτά προκαταλήψεις, στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν. Δυστυχώς ε, ούτε εδώ έχουμε επαρκή δεδομένα ως προς τη διακριτική μεταχείριση κατά των Τούρκων. Το Εθνικό ε, Στατιστικό Ινστιτούτο μας ε, παρακολουθεί τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και 55% των ΡΟΜ παραδείγματος χάρη εξαρτώνται πλήρως από τις κρατικές παροχές αλλά αντίστοιχα ποσοστά δεν έχουμε για τους ΡΟΜ, για τους που έχουν υποστεί διακριτική μεταχείριση, δεν έχουμε καθόλου δεδομένα για την ύπεθρο ε, ή για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ε, στην ύπεθρο. Ξέρουμε ε, ότι υπάρχουν τοκετοί σε χαμηλή ηλικία, 10 έως 15 ετών, και αυτό καταδεικνύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε αυτά τα κορίτσια για τις δυνατότητες που υπάρχουν για τον οικογενειακό προγραμματισμό και την αντισύλληψη. Πριν από 10 χρόνια η Βουλγαρία άρχισε να υλοποιεί ένα πρόγραμμα διαμεσολαβητών για τις υπηρεσίες υγείας, υγείας ε, αυτό μας οδήγησε σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Διοργανώθηκαν ενημερωτικές εκστρατείες ε, για τις εθνοτικές μειονοτικές, ε, για τις μειονοτικές, συγγνώμη, για αυτές τις εθνοτικές ομάδες ε, εργαστήκαμε για να ε, προωθήσουμε την πρόληψη ε, Πλην όμως η προϊόντα διαδικασία μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας προβλέπει τον παροπλισμό διαφόρων νοσοκομιακών μονάδων ε, και υπάρχουν τραγικά ε, περιστατικά όπου τα επίγοντα παραδείγματο χάρη δεν έστειλαν ε, ασθενοφόρα σε γειτονιές όπου μένουν οι Ρώμα ή σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση για να φτάσει το ασθενοφόρο σε αυτά τα χωριά. Ορισμένε φορέ περνάει μια μισή ώρα πριν αποσταλεί και ε, σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που έχω κατά νου, η γυναίκα Ρομ ε, που χρειαζόταν το ασθενοφόρο αποβίωσε πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Είναι ένα ευρύτατο φαινόμενο ε, και υπάρχουν, υπάρχει μια γενική κατακραυγή κατά αυτών των εγκληματικών καθυστερήσεων Έχουμε επίσης ε, διάφορες ε, προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουμε τη διακριτική μεταχείριση στον τομέα της παιδείας, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια. Έχουμε αναλάβει ε, μέτρα για να υλοποιήσουμε μία εθνική σύσταση για την κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης και θα ήθελα να σας δώσω παραδείγματα ε, θετικών ε, εμπειριών στη συνέχεια που είχαμε σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας κύριε Εγιούπ. Λέει η Πρόεδρος, τώρα θα ακούσουμε ε, την κυρία Μπρίτα Τόμψεν για να καταθέσει την προσωπική της μαρτυρία και να μοιραστεί μαζί μας ε, την ανάλυση της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση η οποία με έπεισε ότι υπάρχουν ε, δύο διαφορετικές ομάδες και διαφορετικές ενότητες διότι η, κατάσταση στη Βουλγαρία με την ομάδα των ε, ΡΟΜ είναι διαφορετική και αυτό που βρήκα πολύ ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπατε για την τουρκική μειονότητα στη Βουλγαρία σε σύγκριση με ε, την ε, μειονότητα ΡΟΜ. ποιες είναι οι διακρίσεις τις οποίες υποφέρουν και ε, νομίζω ότι η η είναι ένας ε, από τους ε, πρωταρχικούς ε, ε, λαούς και τα προβλήματα που έχουμε στην ε, Ισλανδία είναι διαφορετικά από αυτά που έχουμε με, με τους Ισλανδούς είναι διαφορετικά αυτά που έχουμε με τους Τούρκους είναι ε, κυνηγοί και ε, τους αντιμετωπίζουμε διαφορετικά πρέπει λοιπόν να γίνει μια τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουν να ενταχθούν οι Ρώμ χρειαζόμαστε πολλές τις στατιστικές και πολλά στοιχεία για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Διότι αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι αυτό το οποίο έγινε ελέγχθη για την εκπαίδευση. Ότι οι άντρες ε, Ρώμ είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι από ό,τι γυναίκες. Βλέπουμε όμως γενικώ σε όλες τις ε, χώρες και στις ομάδες των μεταναστών ότι οι γυναίκες τώρα είναι καλύτερα κατηρτισμένες από ότι οι νέοι. Υπάρχει δηλαδή μία ε, ε, ε, κατάληψη από τις γυναίκες του συστήματος ανωτά της εκπαίδευσης, τουλάχιστον όσον αφορά τις γυναίκες ΡΟΜ. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού σε, πολλά, σε διάφορα νέα κράτη-μέρη ε, και στην Ανατολική Ευρώπη ακούσαμε ε, και άλλους που είπαν ότι το 50% του πληθυσμού, ε, το 15% του πληθυσμού είναι, είναι ρομ. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ε, ένταξη των νεοφερμένων διότι στη δεκαετία του 50 υπήρχαν άτομα από την Νότιο Ευρώπη, από την Ανατολική Ευρώπη, γυναίκες και άντρες. Ενώ τώρα τα, οι θέσεις ε, εργασίες οι οποίες δημιουργούνται και δεν θέλουν να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι είναι στον τομέα των υπηρεσιών. Και καλύπτονται από γυναίκες μετανάστριες στην Ισπανία. Είναι φυσιολογικό η γυναίκα να ε, μεταναστεύσει για 10 μήνες, ε, να μαζέψει χρήματα και μετά να καλέσει τον πατέρα, τον άντρα της ε, και τα παιδιά της για να έρθουν και αυτοί. Ε, η κατάσταση λοιπόν είναι διαφορετική στην Ευρώπη μεταξύ ανδρών και γυναικών και θα αλλάξει ακόμη περισσότερο στο μέλλον διότι οι γυναίκες μπορεί να ζουν σε απόμακρες περιοχές μέσα στην χώρα. Στη Δανία υπάρχουν περισσότεροι ε, άντρε κατά 20% στην Ήπεθρο από ότι στα μεγάλα κέντρα. Άρα η και συγκεντρώνονται στα μεγάλα κέντρα και οι άντρες είναι ικανοποιημένοι να ζουν χωρίς γυναίκες και να παραγγείλουν με το ταχυδρομείο, αυτό που λέμε mail order bride, μία νύφη. Ε, υπάρχουν λοιπόν ε, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου και βλέπουμε ότι οι γυναίκες είτε περιθάλπουν ε, τον γυράσκοντα πληθυσμό ε, ή παντρεύονται με άντρες που δεν μπορούν να βρουν γυναίκα στην περιοχή τους και βλέπουμε τις γυναίκες σε συγκεκριμένα στερεότυπα και με συγκεκριμένο συγκεκριμένη εκπαίδευση ε, όλες ε, λοιπόν αυτές δεν ε, μπορούν να καταστήσουν αποδεκτή την ε, εκπαίδευση που έχουν λάβει. Βλέπω ότι ε, πολλές γυναίκες από τη Μολδαβία, από την Ουκρανία ε, που ήταν για Τρίνες που ήταν δικηγόροι πηγαίνουν στην Πορτογαλία και ε, δουλεύουν ε, για να φροντίζουν ε, ηλικιωμένους. Βλέπετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι εκπαιδευμένες γυναίκες πήγαν να αναλάβουν χαμηλού επίπεδου εργασίες. Ορισμένες κατάφεραν να αντεπεξέλθουν αλλά δεν υπήρχε σύστημα και ίσως το παράδειγμα που αναφέρω είναι πολύ καλό διότι εξετάζει το άτομο. Στη δεκαετία του 60 όταν υπήρχαν άντρες οι οποίοι μετανάστευαν ε, ε, ή στην ε, Γερμανία για συγκεκριμένες δουλειές βλέπουμε ότι τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει, οι γυναίκες έρχονται από διαφορετική προέλευση προσπαθούν όμως να ενταχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω της εργασίας. Οπότε καλύτερα θα πρέπει να κοιτάξει κανείς ποιες είναι οι δεξιότητες του ατόμου, πώς μπορούν να βρουν δουλειά και όχι από πού έρχονται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για να μπορέσει μία ένταξη των ε, συγχρόνων γυναικών και θα ήθελα ε, επίσης να σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό διότι δεν πρέπει μόνο να εξετάσουμε την αγορά εργασίας αλλά πρέπει επίσης να σκεφτούμε πώς οι γυναίκες μπορούν να εμπνευστούν να ασχοληθούν με την πολιτική διότι ε, πρέπει να δούμε πόσο μπορούν να εκλεγούν στην τοπική αυτοδιοίκηση ε, διότι όλοι οι πολίτες της Ευρώπης ε, μπορούν να εκλεγούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και θεωρώ ότι και αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Αυτά όσον αφορά την αναγνώριση. Και η παιδεία είναι βασική για την Ευρώπη. Συνεργαζόμαστε με τη διαδικασία της Μπολόνια και αυτό θα έπρεπε να επεκταθεί και σε περισσότερες χώρες κατά τρόπον ώστε να έρθουν και να εργαστούν εδώ ορισμένοι, διότι τώρα υπάρχει κρίση, υπάρχει ανεργία, αλλά σε λίγα χρόνια θα έχουμε μεγάλες προκλήσεις ελήψεως εργατικού δυναμικού. Και ε, αν δει κανεί τη δημοκρατική κατάσταση στην Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσουμε να εντάξουμε και να αφομοιώσουμε αυτούς τους πληθυσμούς. Σας ευχαριστώ. Έχω όμως και μία ερώτηση ακόμη σχετικά με τη Βουλγαρία και τους Ρομ. Ε, είπατε ότι οι Ρώμο παντρεύονται με, με Τούρκους ή παντρεύονται μόνο ε, με Ρώμ αγοράζουν και, ε, με συγχωρείτε, ε, παντρεύονται και άλλες εθνότητες, Βουλγαρούς, Τούρκους και τα λοιπά ή μόνο Ρώμ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τόμσεν. Κατόπιν αυτού θα ξεκινήσω τώρα τη συζήτηση και είμαι στη διάθεσή σας να συγκεντρώσω τις ερωτήσεις καταρχήν από τις ευρωβουλευτίνες που είναι στην αίθουσα και χαιρετίζω την κυρία Ρόδη Κράτσα που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ήρθε. Ε, άρα η κυρία Κράτσα πρώτα και ε, της δίνω το λόγο σε αυτό το θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ και είναι πολύ βασικό για μας στην ευρωπαϊκή μας κοινωνία εδώ σήμερα. Κυρία Πρόεδρε, ε, ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτής της ε, δημόσιας ακρόασης σήμερα και να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους, τους ειδικού που ήλθαν να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες τους. Θέλω να πω ότι το θέμα που σήμερα μας απασχολεί είναι πολύ σημαντικό ε, και για την εσωτερική συνοχή και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια κοινωνία με πλήρη απασχόληση, με συνοχή, με κοινωνική ειρήνη, με ευημερία, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για την πολιτική γειτονία και για την πολιτική των εξωτερικών σχέσεων. Διότι η, η, είναι αλληλένδετα η εσωτερική κατάσταση, η συνοχή, η ασφάλεια με την πολιτική που έχουμε για την ε, ανάπτυξη στις χώρες που είναι γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι υποψήφιες χώρες, είτε είναι χώρες ε, εταίροι, ε, και βέβαια και για τις χώρες που βρίσκονται ακόμη πιο μακριά και οι οποίες είναι χώρες προέλευσης μεταναστών. Λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι όλα τα θέματα τίθενται στο τραπέζι, όλες οι εθνοτικές ομάδες. Ε, και θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και για τα μέλη της Επιτροπής, τα καινούργια ίσως μέλη της Επιτροπής, αλλά και για τους εμπειρογνώμονες που θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθειά μας, ε, να βασιστούμε και στα κείμενα που έχει ήδη ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εκθέσεις που έχει κάνει για τις γυναίκα Ρώμα, για τις γυναίκες ε, μετανάστριες, διότι το, το ακεί, τα δεδομένα Α της Επιτροπής μας είναι πολύ σημαντικά, διότι το Κοινοβούλιο έχει συνέχεια και είναι πολύ σημαντικό να βασιστούμε σε παλαιότερα κείμενα και ψηφίσματα, να δούμε τι από αυτά έχουν υλοποιηθεί, γιατί δεν έχουν υλοποιηθεί και τι καινούριο μπορούμε να δώσουμε. Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη προσφορά που κάνουμε και στην πολιτική μας πράξη, αλλά και στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε και μένα να εκφράσω την άποψή μου. Σας ευχαριστώ. Merci, ευχαριστούμε, κυρία Κράτσα. Η κυρία Ένς τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σκέφτηκα ε, αν θέλουμε να καταρτήσουμε μία στρατηγική κατά των διακρίσεων για τις γυναίκες διαφόρων εθνοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει μία, ένα σαφής διαχωρισμός για το θέμα που συζητάμε δηλαδή πότε μετανάστευσαν οι γυναίκες, γιατί μπορεί να είναι τελείως διαφορετικές γενιές. Ε, τι έχει συμβεί με την παλιά γενιά, τη νέα γενιά, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειας και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δυσχερές. Αλλά οι μουσουλμάνες γυναίκες είναι ένα διαφορετικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί χωριστά. Και αυτή η ποικιλία των προβλημάτων των ε, ε, μειονοτήτων, διαφόρων εθνοτήτων πρέπει να εξεταστούν για να επιτύχουμε και να καταργήσουμε τις διακρίσεις σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε και να συμβάλλουν και τα κράτη-μέλη. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, ποιες είναι οι, διαφορετικές, οι διαφορές πρέπει να ληφθούν υπόψη και ποια είναι τα κοινά στοιχεία και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, διότι αυτό είναι το βασικό μας ερώτημα, να ακούσω κάποια λύση από τους προσκεκλημένους μας. Δηλαδή, εσείς ποια θεωρείτε ότι είναι τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν, από πού έρχονται οι γυναίκες, ποιες είναι οι γενικές γραμμές τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ίσως κάτι μπορείτε να μας πείτε του θέματος αυτού. Ευχαριστώ, η κυρία Κιλ Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εφόσον μιλάμε για έλλειψη δεδομένων, ε, εγώ ε, σκέφτηκα τις ε, Αυγανές γυναίκες ε, που κρύβονται πίσω από την μπουρκα δεν υπάρχουν μπουρκες στην Ανατολική Ευρώπη αλλά δεν βλέπουμε αυτές τις γυναίκες είναι κρυμμένες πρέπει να αναφερθούμε επίσης στα στατιστικά δεδομένα διότι αυτό είναι πολύ βασικό αν θέλουμε όντως να δούμε την κατάσταση και είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει, δηλαδή να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίες οι γυναίκες αυτές μετανάστευσαν. Πρέπει να τεθεί το βασικό ερώτημα γιατί κάποιος λαός βρίσκεται στην Ευρώπη και πώς μπορούμε να απαντήσουμε ε, να βρούμε τους λόγους και τις αιτίες ε, συνολικά της ε, μετανάστευσης διότι υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει εφόσον φυστάμεθα την μετανάστευση. Όσον αφορά τη δικιά μου περιοχή εγώ ζω ε, ε, δυτικά αλλά στο βορρά υπάρχουν πολλοί ε, Ρομ στη Γαλλία και ε, το ερώτημα που πρέπει να τεθούμε είναι γιατί είναι τα άτομα αυτά, γιατί έχουν μεταναστεύσει, γιατί βρίσκονται εδώ, γιατί βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης. Επέλεξαν να μείνουν εκεί ή υφίστανται, γιατί υφίστανται αυτή την ε, μετανάστευση και πώς μπορούμε εμείς υπό αυτές τις συνθήκες να επέμβουμε στις αιτίες αυτού της μετανάστευσης. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, ο κύριος Φωτάκης, θέλετε να κάνετε μία ερώτηση. Θα ήθελα καταρχήν να επέμβω σχετικά με αυτό το οποίο είπε η κυρία Ένστ. Γιατί αισθάνομαι ότι είμαι εμπειρογνώμων σε δημογραφικά θέματα και μετά θέλω να απευθύνω και μία ερώτηση. Καταρχήν, πολλές φορές ε, ε, δραματικοποιούμε ε, το δημογραφικό θέμα διότι θεωρούμε ότι έχουμε ανάγκες που δεν θα καλυφθούν. Πιστεύω όμως ότι μετά τα δύο χρόνια της οικονομικής κρίσης η κατάσταση είναι τέτοια ώστε το πιο πιθανό σενάριο για την επόμενη δεκαετία είναι ότι θα έχουμε ε, και ε, ανεργία και ανικανοποίητους ε, εκπαιδευμένους εργαζομένους διότι υπάρχει μία δομή. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε την οικονομία μας στις νέες πραγματικότητες. Βλέπουμε ε, ήδη ε, θέματα ε, όσον αφορά την συνεργασία παραδείγματος χάρη μεταξύ της Ρενό και της Ντέμπλερ εχθές. Ε, στα θέματα λοιπόν αυτά και στο περιβάλλον αυτό θα χρειαστούμε νέες δεξιότητες και έχουμε ε, ένα σωρό άτομα που χάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι εύκολο να πάρουμε τους ανέργους αυτούς και να τους χρησιμοποιήσουμε για τις νέες δεξιότητες. Δημογραφικά λοιπόν λοιπόν όλα τα οι νεοφερμένοι και νεοεκπαιδευμένοι με νέες δεξιότητες δεν επαρκούν γιατί η νέα γενιά είναι πολύ μικρή, πολύ πιο περιορισμένη πρέπει να καλύψουμε το κενό λοιπόν με μετανάστες και αυτό είναι το βασικό θέμα που θα μας απασχολήσει την επόμενη δεκαετία δηλαδή μετά θα χρειαστούμε και μαζικά ανάγκες σε εκπαιδευμένο προσωπικό για 45 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν μία τάση αλλά με διαφορετικές φάσεις. Ε, τώρα, έχω να κάνω μία προκλητική ερώτηση. Όταν μιλάμε για ένταξη, το πρώτο που λέμε πάντοτε είναι ότι η ένταξη αναφέρεται και στην κοινωνία που υποδέχεται και στους μετανάστες. Όταν όμως μιλάμε για μέτρα, εμείς μιλάμε για μέτρα που απευθύνονται στους μετανάστες και όχι στην ε, την κοινωνία που φιλοξενεί. Δηλαδή, ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την κοινωνία που θα υποδεχθεί τους μετανάστες. Διότι το βασικό παράπονο των μεταναστών είναι ότι ακόμη ε, και αν ε, χαίρονται ε, για τις ενέργειες που γίνονται υπέρ αυτών, αυτό γίνεται σε ένα κενό. Μαθαίνουν τη γλώσσα αλλά δεν έχουν επαφή με τη γλώσσα. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω λοιπόν είναι αν υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές που να απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία. Ευχαριστώ κύριε Φωτάκη. Επαναρχόμαστε λοιπόν στην εμπειρία που μας περιέγραψε η κυρία Μέλλερ Γιάνσεν η οποία μίλησε ε, για τον ε, επαγγελματισμό της ε, και όπως είπε και η κυρία Κράτσα προηγουμένως θα πρέπει ε, να διαχωρίσουμε ε, το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ της υποδοχής και των μεταναστών ε, και να ασχοληθούμε με τις αξίες που διαμορφώνουν την κοινωνία μας. Το δεύτερο πολύ βασικό θέμα που μας ε, έθιξε ο κύριος Σεγιούπ είναι ότι έχουμε έλλειψη δεδομένων όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ του προβλήματος της ε, ε, κοινωνικής εντάξεως μεταξύ υπαίθρου και αστικών κέντρων. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι οι εμπειρία που έχετε σε αυτό το τομέα. Κυρία Μέλλερ Γιάνσεν, έχετε καταρχήν το λόγο για να, μιλή, για να απαντήσετε στο πρώτο μέρος των ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω πως ε, πέρσι τον Νοέμβριο διοργανώσαμε μια διεθνή διάσκεψη υπάρχουν τα πάντα στα, στα αγγλικά, οι ιστορίες των ζευγαριών εκεί πέρα στην ε, σελίδα μας kvinfo.dk ε, υπάρχουν πολλές φιλοφορίες εκεί Τώρα για τα θέματα των δεδομένων. Όλα αυτά τα χρόνια τα αποτελέσματα των ε, συνεντεύξεών μας με τους μέντορες ε, και αυτούς που βοηθούσαν τα βάζαμε στην βάση δεδομένων. Αλλά στην αρχή δεν ξέραμε πόσο μεγάλο θα γινόταν αυτό το πρόγραμμα Οπότε ήταν ε, μόνο ένα εργαλείο εσωτερικό. Αλλά τώρα αναπτύσσουμε αυτή την βάση δεδομένων ε, για να μπορέσουμε να βρούμε τις απαντήσεις, ποιοι προέρχονται δηλαδή από ποια χώρα, τι εκπαίδευση έχουν για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε αποτελέσματα. Οπότε σε έξι μήνες θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί βεβαίως είναι μοναδικό το υλικό. Δεν νομίζω πως κανείς άλλος έχει αποτελέσματα έξι ετών ε, παρακολούθησης αυτών των γυναικών. Και ε, κάποιος ρώτησε για την δεκαετία του του Για, με συγχωρείτε για τις ηλικίε. Οι ηλικίε είναι όσον αφορά τους μέντορες μεταξύ 25 και 55. Η πλούσια είναι γύρω εκεί στα, στα 35. Οπότε και για τις κοινωνίες και για την οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενσωματωθούν αυτές οι γυναίκες. Δεν ξέρω τώρα η Γερμανίδα κυρία με ρώτησε, μου ζήτησε να κάνω μια διάκριση μεταξύ των διαφόρων ομάδων από που προέρχονται δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κινητοποιηθεί λοιπόν η κοινωνία των πολιτών και γι' αυτό πρέπει να μην κάνουμε διάκριση, δηλαδή από πού προέρχεται ο καθένας, εάν είναι μουσουλμάνος αλλά να δώσουμε βάρος, να εστιάσουμε στα άτομα. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω πω για έναν πολιτικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασιστική σημασία το να μπορεί να κάνει αυτή την διάκριση, αλλά νομίζω πως η μέθοδος μας είναι τμήμα της επιτυχίας μας, ότι ακριβώς δεν το κάνουμε αυτό, γιατί εγώ θέλω να ανοίξει ακριβώς ε, το Ίδρυμά μας και για τις ε, νέες γυναίκες, τις μουσουλμάνες, να μην ε, θεωρούνται μουσουλμάνες κατά κύριο λόγο. Τις προσκαλούμε στο πρόγραμμα αυτό, στο Ίδρυμα, ως άτομα με το δυναμικό που έχουν, με τις ελπίδες τους, με όλους τους πόρους που έχουν. Τους προσκαλούμε λοιπόν να ενταχθούν, ε, τους δίνουμε μία ορμή για να γίνουν τελικά Δανέζες, να αποτελέσουν τμήμα αυτής της χώρας. Οπότε υπάρχει το θέμα αυτό της κινητοποίησης της κοινωνίας των ε, πολιτών, αλλά είναι βεβαίω οι δικές σας ανάγκες διαφορετικές. Θέλετε να υπάρξει μια ανάλυση. Δεν ξέρω αν σας αρκούν αυτά για την ώρα. Σας ευχαριστούμε, ο κύριος Γιούπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απαντήσω στις ερωτήσεις κυρίας Τόμσεν. Στη Βουλγαρία και η Ρώμα και οι Τούρκοι δεν είναι απαραίτητα μετανάστες. Οι Τούρκοι ε, εδώ και 600 χρόνια μένουν στη χώρα μας, η Ρώμα ακόμη περισσότερο. Και άρα ε, για να ενταχθούν θα πρέπει να θεσπιστεί μια στοχευμένη ε, κυβερνητική πολιτική στη Βουλγαρία. Έχουμε πάρα πολλά θετικά βιώματα. Ε, δυστυχώς όμως υπάρχουν περισσότερες αρνητικές εμπειρίες λόγω των προκαταλήψεων που οδηγούν στις διακρίσεις. Για να αποφευθούν οι διακρίσεις θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στη φροντίδα των παιδιών ήδη από τον υπηαγωγείο για να εγγυηθούμε την εκπαίδευσή τους ε, μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι, αυτές οι ελλείψεις οδηγούν ε, στην άρνηση των ΡΟΜ από την ε, κοινωνία. Πολύ συχνά οι νέοι μέσα στις ε, τάξεις δεν θέλουν κάτω στο ίδιο θρανείο με ένα παιδί ρομ. Διαπιστώνεται λοιπόν αυτή η διακριτική μεταχείριση κατά και των ανάπηρων παιδιών. Ε, οι Ρομ συνήθως ε, παντρεύονται Ρομ. Μικτή γάμη, η μεικτή γάμη είναι ολγάριθμη στη, στη Βουλγαρία. Θα σας δώσω ένα τραγικό παράδειγμα, κάτι που συνέβη πριν από 5-6 μήνες. Υπήρχαν δύο ερωτευμένοι, φανταστείτε τον Ρωμαίο και, τον, και την Ιουλιέτα, 6-7 χρονών, εκείνη ε, Βουλγαρία, εκείνος ε, Ρώμ, ε, λοιπόν αυτοκτόνησαν, έπεσαν στις γραμμές του τρένου, το κοριτσάκι πέθανε, ενώ το αγόρι ακροτηριάστηκε. και ε, ε, ε, προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν λόγω του κοινωνικού στιγματισμού, διότι λόγω των προκαταλήψεων δεν μπορούσαν να είναι μαζί. Ε, επίσης, μην ξεχνάμε ότι είμαστε μεθοριακή χώρα στο χώρο του Σέγγεν και υπήρχαν φόβοι ότι θα έχουμε μαζική εισρωή Ρώμα στις δυτικές χώρες. Ε, τελικά όμως ε, διαψεύστηκαν αυτοί οι φόβοι. Αλλά ε, πρέπει να διερευνήσουμε, να εξηχνιάσουμε για ποιους λόγους μεταναστεύουν οι Ρώμ. Τις περισσότερες φορές είναι για να εργαστούν κάπου. Και οι, οι περισσότεροι Ρώμ είναι γυναίκες, Δηλαδή οι άντρε δρομένουν στο σπίτι για να φροντίσουν τα παιδιά και βγαίνουν να δουλέψουν οι γυναίκες. Και τώρα προσπαθούμε να ε, κινητοποιήσουμε τους ε, Ρώμες στη Βουλγαρία για να επιτύχουν τη χειραφέτηση των ε, γυναικών. Τώρα για την διαφορά ανάμεσα στις αστικές ζώνες και την Ήπεθρο. Λοιπόν, στην ε, Ήπεθρο είναι ευχερέστερη η ένταξη, γιατί γνωρίζουν οι μεν τους δε και δεν ε, υπάρχει τόσο μεγάλη διάκριση ούτε σε επίπεδο γειτονιάς, ούτε σε επίπεδο σχολείου. Το πρόβλημα είναι ε, βιοποριστικό και επίσης ε, το, υπάρχει το πρόβλημα της ε, αστιφιλίας λόγω της οποίας ε, κλείνουν νοσοκομεία, κλείνουν σχολεία στα χωριά και διωγγώνονται τα προβλήματα που τόσοι ή υπάρχουν στις πόλεις. Θα ήθελα να προσθέσω ότι στην Βουλγαρία δεν υπάρχουν ομάδες ρομ, δεν πρόκειται για οδηπόρους, για ρομ που ταξιδεύουν. Έχουν καθιστική θα έλεγα ζωή, επιλέγουν ε, εγκαθίστανται σε μια συγκεκριμένη περιοχή έχουν πρόσβαση στην αποχέτευση, στην ηλεκτροδότηση κτλ. Αλλά το πρόβλημα είναι ο υπερπληθυσμός μέσα σε αυτές τις συνοικίες ΡΟΜ. Συχνά οι ΡΟΜ επίσης ε, κατασκευάζουν ε, Παραγκούπολης, ε, Παραγκούπολη, συγγνώμη, ή άλλους πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς κανένα σχέδιο πόλης φυσικά, χωρίς καμία άδεια πολεοδομίας. Και γι' αυτό σας εξηγούσα προηγουμένως ε, ότι ε, είναι απαραίτητο να έχουμε στατιστικά στοιχεία, να ξέρουμε πόσα παιδιά τελικά πηγαίνουν στο σχολείο, πόσοι μένουν στο σπίτι, πόσοι είναι στην αγορά εργασίας, ε, πόσοι είναι οι μη δηλωμένοι άνεργοι, διαφόρων ειδών στατιστικά δεδομένα που θα μας επιτρέψουν τελικά να λύσουμε το πρόβλημα. Ε, ε, αν δεν έχουμε δεδομένα δεν μπορούμε και να αναλάβουμε κανένα μέτρο. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιούπ για τις απαντήσεις που μας δώσατε, λέει η Πρόεδρος. Κλείνει τώρα το δεύτερο πάνελ για τις πρακτικές ως προς την ένταξη και θα περάσουμε στο τρίτο τμήμα τώρα της ε, σημερινής μας με κάποιες ε, εισηγήσει για μέτρα, συγκεκριμένες προτάσεις. Ε. Θα ακούσουμε την κυρία Άμαντιν Μπάκα από το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών ε, που ήρθε εδώ στο βήμα και κατόπιν ε, την κυρία Μπάουερ και την κυρία Κιλ Νίλσεν. Παρακαλώ. Thanks. Um, I would like first to... ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την Επιτροπή Γυναικών ε, και την εισηγήτρια της έκθεσης, την κυρία Παρβάνοβα που μας κάλεσε αν και είναι έκθεση ίδιας ε, πρωτοβουλίας και επειδή ακούσαμε πάρα πολλές προτάσεις πολιτικής ε, από το πρωί, εγώ θεωρώ πως είναι καθήκον μου να επισημώνω κάποιες προτάσεις που σχετίζονται άμεσα με κάποιες συζητήσεις που γίνονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ακούσαμε αρκετές προτάσεις και δεν πρέπει να τις ε, ξεχάσουμε και Εκεί θα κάνω την σύνδεση με τα τρέχοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κάνω λοιπόν την σύνδεση όταν μιλάω για τα τρέχοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που θα επηρεάσει τις μειονοτικές γυναίκες αναφέρομαι στη στρατηγική του 2020 που θα παίξει ένα ρόλο κλειδί στην ενσωμάτωση αυτών των γυναικών. Αναφέρομαι στη νέα στρατηγική ισότητα των φύλων που συζητιέται αυτή τη στιγμή. Και νομίζω σήμερα στις 5 οι τροπολογίες ε, της έκθεσης ε, της Επιτροπής Γυναικών θα κατατεθούν το σχέδιο δράσης ε, του προγράμματος Στοκχόλμης όταν μιλάμε για τις μετανάστριες θα έχει και αυτό τη σημασία του. Η ενσωμάτωση είναι ευθύνη των κρατών μελών, αλλά με την συνθήκη της ε, Λισαβόνας είναι, υπάρχει ένας διαφορετικός μηχανισμός. Οπότε σιγά σιγά είναι υπόθεση και της Ένωσης και η Κομισιόν και η Ένωση έχει μεγάλο ρόλο να παίξει. Έχουμε τις κοινέ βασικές αρχές, ε, τις οποίες αναφερθήκαμε σήμερα το πρωί όταν μιλήσαμε για την ε, διμερή διαδικασία και αυτά τα ξεχνάμε. Τα συζητήσαμε λοιπόν σήμερα το πρωί και η ευθύνη είναι στις μετανάστριες. Μιλάμε για μαθήματα γλώσσας και ξεχνάμε πως είναι και η κοινωνία υποδοχής. Ε, το είπε και ο κύριος Φωτάκης. Γιατί δεν έχουμε δείκτες για το πώς η κοινωνία υποδοχής αυτό είναι σημαντικό και είναι κάτι που ξεχνάμε συχνά γιατί αποτελεί ενσωμάτωση ένα μέσο πολιτικής και καμιά φορά πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω, να ακούσουμε όπως κάναμε σήμερα το πρωί τις φωνές ε, στο επίπεδο των ανθρώπων που βλέπουν το αντίκτυπο αυτών των πολιτικών στις ζωές ε, των ε, μεταναστριών, των γυναικών Ρωμά, των διαφόρων μειονοτήτων. Πριν προχωρήσω παραπέρα, να εξηγήσω κάποια πράγματα. Οι περισσότεροι γνωρίζετε ποιο είναι το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών. Είμαστε μεγαλύτερη οργάνωση συνδέσμων γυναικών με πάνω από 2.500 μέλη, οργανισμούς μέλη. Βασιζόμαστε στα μέλη μας και όπως είπα και στην αρχή ε, δίνουμε βάρος στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά έχουμε και δραστηριότητε σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Στη δουλειά μας, εγώ ε, εργάζομαι στην ενσωμάτωση, άσυλο, κατά καταπολέμηση των διακρίσεων, αλλά έχω συναδέλφου που εργάζονται στις κοινωτικές πολιτικές, γυναίκες στη λήψη αποφάσεων, διακατά των γυναικών ευρωπαϊκές πολιτικές και νομοθεσία ισότητας. Όλα αυτά τα θέματα νομίζω βεβαίως άμεσα σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των μειονοτικών γυναικών και θα προσπαθήσω όπως σας είπα να αναφερθώ συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικές και όχι μόνο στην καταπολέμηση των διακρίσεων και τη μετανάστευση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για τη δουλειά που κάνουμε. Πρόσφατα είχαμε μια δημοσίευση, την έχω βάλει εκεί μπροστά στην είσοδο, για την καταπολέμηση των διακρίσεων και εξετάζει συγκεκριμένα την, το που συναντιόνται διάφορα είδη διακρίσεων, π.χ. φίλο και φιλή. Υπάρχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας για τις διακρίσεις που λέγεται Φίλο και Φιλή και μην ξεχνάτε μπορείτε να επηρεάσετε την έρευνα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα άρθρο λοιπόν εδώ πέρα και εμείς ε, το σχεδιάσαμε αυτό για, ως ένα πρακτικό εργαλείο για όλους είτε εργάζονται στην καταπολέμηση των διακρίσεων ή την ισότητα πιο συγκεκριμένα για να δουν ε, την ε, σύνδεση. Ένα άλλο έργο που κάνουμε παράλληλα το οποίο χρηματοδότησε το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων είναι να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου δικτύου μεταναστριών και πρόεδρος βεβαίως είναι η Βερτζίνια που σας μίλησε το πρωί γιατί είναι σημαντικό σας ευχαριστούμε γι' αυτό οι φωνές αυτών που ξέρουν την πραγματικότητα να ακουστούν απευθείας στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να μπορέσουν αυτοί που ασκούν την πολιτική να ακούσουν αυτούς απευθείας και όχι εμάς τους ενδιάμεσους. Ένα από τα βασικά ζητήματα και αυτό θα σας ζητήσω σήμερα είναι πως ο καθένας από εμάς όπου και αν βρίσκεται, είτε είναι στο ευρωπαϊκό επίπεδο και δουλεύει για την Κομισιόν, είτε είναι ευρωβουλευτής, είτε δουλεύει σε κάποια μικιό, να έχει μία προοπτική έτσι, η οποία θα είναι τομή μεταξύ διαφόρων τομέων. Και βεβαίω συχνά ακούγεται αυτή η λέξη χωρί να ξέρουμε το τι σημαίνει στην πράξη. Θα κάνω λοιπόν κάποιε συγκεκριμένε προτάσει για το πώ θα μεταφερθεί στην πράξη. Το ανέφερε νομίζω η Ισαμπέλα στην ομιλία τη, καθώ υπάρχει διακριτική μεταχείριση με βάση το φύλλο, αν και συχνά υπάρχουν παρόμοιε διακρίσει όταν μιλάμε π.χ. για τη στέγαση αυτών των γυναικών Ρωμά υπάρχουν διαφορετικές διακρίσεις γιατί είσαι και γυναίκα ε, και Ρωμά, γιατί είσαι και μαύρη και γυναίκα. Ε, σε κάποιες χώρες όπου επιτρέπονται τα εθνοτικά στοιχεία όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ενδιαφέρουσα έρευνα για, το, για την απασχόληση των μαύρων γυναικών π.χ. Και εκεί πέρα βλέπουμε την πολλαπλή διάκριση που υφίστανται έχω τονίσει διαφορετικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου είναι σημαντικό να εργαστούμε με μια τέτοια κοινή προσέγγιση, γιατί συχνά ε, ασχολούμαστε με τις μετανάστριες, αλλά ξεχνάμε πως καμιά φορά χρειαζόμαστε στοχευμένες πολιτικές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ κοίταξα παραδείγματος χάρη αυτό τον οδικό χάρτη, την έκθεση που συζητιέται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω πως μια τέτοια ισχυρότερη προοπτική θα ήταν χρήσιμη σε αυτή την έκθεση. Π.χ. οι γυναίκες θα επωφελούνταν από αυτό το σχέδιο ισότητας. Αυτή ήταν η θέση μας και πέρσι. Τα, θα μπορείτε να τα δείτε αυτά και στη σελίδα μας. Επίσης, ε, καλωσορίζω την παρέμβαση της ε, κυρίας Καράτσα όταν ε, υπενθύμησε πως δεν είμαστε σε ένα κενό πολιτικής. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε την, και τη σύμβαση του 1979, είναι πάνω από 30 χρόνια, 30 χρόνια ήταν πέρσι, και έχουμε και την οδηγία ισότητας ε, φιλετικής ισότητας, αλλά βλέπουμε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο πληθαίνουν οι φωνές για να δώσουμε προσοχή συγκεκριμένες ομάδες γυναικών, είτε είναι Ρωμά, μετανάστριες, μειονοτικές γενικότερα. Και εγώ ανέφερα και το ψήφισμα για τις ε, Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο τόνισε η Κιζαμπέλα, που υπήρχαν γυναίκες και υπήρχαν δεδομένα αναλυμένα ανά ε, εθνότητα και φίλο και είχαν γίνει κάποιες πάρα πολύ καλές στάσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Το ψήφισμα για τη μετανάστευση των γυναικών που ανέφερε η κυρία Κράτσα που είχε συνταχθεί τότε. Χρήσιμη έκθεση και έκθεση της Ζαμπέλας για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Υπάρχει επίσης μια προοπτική Φίλου στην νομοθεσία περί διακρίσεων. Εκεί λοιπόν που υπάρχουν διαφορετικές ομάδες και είναι π.χ. Ρωμά, Μουσουλμάνοι, άντρες γυναίκες, δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι καταγγελίες γιατί δεν εμπιστεύονται, δεν ξέρουν κιόλας και ειδικά οι Ρώμα ξέρουν, αλλά δεν εμπιστεύονται τους φορείς στους οποίους πρέπει να κάνουν καταγγελίες. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις πολιτικής για να το αλλάξουμε. Και αυτό νομίζω ε, είναι και ένα από αυτά τα οποία είπαμε σήμερα το πρωί. Έχουμε δέσμευση, έχουμε πάρα πολλές δεσμεύσεις ε, ε, λέγεται το πώς πρέπει να δώσουμε βάση σε συγκεκριμένες ομάδες. Τώρα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Δράσεις, συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Η Βιρτζίνια επίσης αναέφερε στην ομιλία της τι πρέπει να κάνουμε. Ήταν πολύ λεπτομερές αυτό το οποίο είπε. Πρέπει να μειωθεί ο χρόνος που περιμένουν οι γυναίκες οι γυναίκες για να ε, αποκτήσουν καθεστώς ε, κατοίκου. Αναφέρθηκε αυτό νομίζω και στην έκθεση Κράτσα που υπεψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει δηλαδή να περάσουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Γιατί ε, ο διάβολος ορισμένες φορές κρύβεται τις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές, αλλιώς λέμε συνεχώς, κάνουμε γενικές δηλώσεις οι οποίε καλέ είναι, ήταν επίτευγμα να γίνουν αυτέ τι δηλώσει, αλλά πρέπει να πάμε τώρα παραπέρα. Μιλήσαμε επίση για τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα και δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτό τα οποία ακούστηκαν. Είναι ουσιαστικό αυτό, αλλά έχουμε ήδη πολλέ ποιοτικέ έρευνε και ποσοτικές και δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Πρέπει να τις αναπτύσσουμε συνεχώς, ειδικά όταν συλλέγουμε δεδομένα για το άρθρο 19 π.χ. τώρα της ε, συνθήκης για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε ήδη αρκετές ποιοτικές έρευνες, υπάρχει έρευνα για την απασχόληση των μεταναστριών που χρηματοδότησε η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Πρέπει λοιπόν να τη χρησιμοποιήσουμε. Χρηματοδότηση, χρηματοδότηση, χρηματοδότηση λοιπόν. Χρειαζόμαστε λεφτά πρώτα απ' όλα για τι πολιτικές. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε καιρού οικονομική κρίση. Πρέπει να αναφερθεί και η οικονομική κρίση. Είναι ουσιαστικό. Χρηματοδότηση επίση, αυτό είναι κοινό νομίζω, για τι μειονοτικές γυναίκε και τι μετανάστριες και τι οργανώσει του, γιατί η χρηματοδότηση ε, είναι δύσκολη. Τότε θα απευθύνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς έχετε ρόλο στον προϋπολογισμό της κοινότητας, να δώσετε τη δυνατότητα σε όλες αυτές τις ομάδες των γυναικών να έχουν πρόσβαση στη, στην κοινωτική χρηματοδότηση για να οργανώσουν εκπαίδευση, να μην έχουν τόσες απαιτήσει χρηματοδότηση έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση υπήρξε μια αξιολόγηση του Ταμείου Ενσωμάτωσης. Μόνο 2% των οργανώσεων ήταν εταίροι στο πρόγραμμα αυτό και έχουμε ένα 70% μήκυο και κανείς δεν είναι ηγέτης, μόνο διάδοση αποτελεσμάτων και δικαιούχοι. Για να ολοκληρώσω κάποιες ε, συστάσεις για την διάκριση Μιλήσαμε για την πολλαπλή διάκριση, μια ρήτρα που πρέπει να συμπεριληφθεί στην εθνική νομοθεσία. Καλωσορίσαμε τη συμπερίληψη αυτής της ρήτρα στην ε, περσινή έκθεση του Κοινοβουλίου με τη νέα οδηγία Κατά πολέμηση των διακρίσεων. Δεν είναι στις συζητήσεις του Συμβουλίου γιατί είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα και ελπίζουμε πως η οδηγία θα υιοθετηθεί. Η απασχόληση το ανέφερα ήδη το είπαμε σήμερα το πρωί, δεν θα πω τίποτα άλλο. Επανένωση οικογενειών. Η Βιρτζίνια το ανέφερε. Είναι ουσιαστικό. Θα γίνει συζήτηση για την επανένωση οικογενειών γιατί η Κομισιόν θα εκδώσει μια πράσινη βίβλα οπότε εσείς ως Ευρωβουλευτές στη συζήτηση αυτή πρέπει να φροντίσετε να μην υπάρχει διάκριση φύλου όταν μιλάμε για την επανένωση οικογενειών, καθώς η τάση που υπάρχει στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να αυξηθούν τα εμπόδια, οι οι περιορισμοί. Άσυλο. πολύ από την ομοθεσία ασύλου εμποδίζει την ενσωμάτωση των γυναικών όταν δεν έχουν το δικαίωμα να εργαστούν. Όταν είναι υποχρεωμένε να ζουν σε απομακρυσμένε περιοχές όπου είναι κάποιο στιγματισμένος, κάποια στιγματισμένη γιατί είναι μαύρη. Έχω κάποια εμπειρία π.χ. και από την, στην, στην Ιλλανδία. Βία θα τελειώσαμε αυτό. Αυτό είναι κρίσιμο για την ένταξη των μεταναστριών. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ε, όσον αφορά το στίγμα. Η βία κατά των γυναικών ε, αφορά όλες τις ομάδες. Υπ' αυτή την έννοια δηλαδή υπάρχει και στην έκθεση Ταραμπέλα. Ζητούμε μια οδηγία για τη βία κατά των γυναικών και ένα συνολικό σχέδιο δράση. Τώρα πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να παίξει έναν ηγετικό ρόλο εδώ πέρα και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τις μετανάστριες. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ κυρία Μπάχ για τον τρόπο με τον οποίο ε, μας υπενθυμίσατε ιδίω τα θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φωτάκη που φεύγει και τώρα δίνω τον λόγο στην κυρία Έντις Μπάουερ για να μας παρουσιάσει την ανάλυση της κατάστασης σχετικά με τα μέτρα που είναι εφικτά και διαθέσιμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτή τη συζήτηση εύκολα. Θέλω να πω ότι ε, θαυμάζω το θάρρος της κυρίας Παρβάνοβα που άνοιξε αυτό το θέμα διότι όπως είπε και η κυρία Γιανακουδάκη δεν υπάρχει ε, καν δεσμευτικός ορισμός των ε, μηνιονοτήτων, των εθνοτήτων από εθνότητες και θα ήθελα να αναφέρω τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης που περιλαμβάνει έναν τέτοιον ορισμό των εθνοτικών μειονοτήτων και εφόσον δεν υπάρχει άλλος πιο δόκιμος ορισμός θα ήθελα να πω ότι χρησιμοποιείται σε ορισμένα έγγραφα όπως η ε, σύμβαση του Φράιμπουργκ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης των Περιφερειακών και μειωνοτικών γλωσσών. Υπάρχουν πέντε χαρακτηριστικά εθνικών μειονοτήτων να διαμένουν ε, στα κράτη και να είναι ε, πολίτες των κρατών αυτών. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει σχετικά με την ε, ρωσική μειονότητα εις τις χώρες της Βλαστικής, και είναι κάτι που θέλω να σας υπενθυμίσω να υπάρχουν σταθερές ε, σχέσεις διαρκείας με το κράτος, ε, ε, χαρακτηριστικά γλωσσικά, πολιτιστικά και παραδοσιακά που διαχωρίζουν από τον υπόλοιπο πληθυσμό του κράτους ή της περιοχής και να υποκινούνται από ενδιαφέροντα που καθορίζουν την εθνική τους ταυτότητα, θρησκεία και ιδιότητες. Παρόλα αυτά, εφόσον υπάρχει κάποιος ορισμός θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία και η Ελλάδα δεν δέχονται στην νομοθεσία τους, δεν αναγνωρίζουν τις μειονότητες. Στο Βέλγιο είναι διαφορετική η κατάσταση, ε, αναγνωρίζουν τις εθνικές μειονότητες αλλά όχι τις, ε, ε, τις εθνικές κοινότητες αλλά όχι τις μειονότητες. Ε, όλα αυτά δεν οριοθετούνται εις την σύμβαση πλαίσιο για τις μειονότητες και όλα αυτά μας αποδεικνύουν ότι μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Αφενός τις εθνικές μειονότητες και ε, την, ε, ε, τους μετανάστες που είναι δύο διαφορετικά θέματα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση Μωράης το 2005 σχετικά με την προστασία των ε, μειονοτήτων και των ε, ε, πολιτικών ενάντια της διακρίσεις στην Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει μία σαφή διάκριση μεταξύ των κοινοτήτων ΡΟΜ των εγκατεστημένων μειονοτήτων, των γλωσσικών των μειονοτήτων, των ε, ε, ε, απατρίδων και των ατόμων που είναι εγκατεστημένα σε μία περιοχή. Διότι αυτές είναι, αυτά είναι τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις μειονότητες και δεν μπορούμε συλλήβδη να διατυπώσουμε μία πολιτική ή μία σύσταση ε, που ε, να ε, μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικές μειονότητες. Έχοντας όμως υπόψη τα στοιχεία αυτά, δεν είναι εύκολο να βρούμε την σωστή σύσταση διότι οι διάφορες μειονότητες ζουν σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Δεν μπορεί να συγκρίνει κανείς την φιλανδική μειονότητα ή ε, την Σουηδία ή την ε, Ουγγρική μειονότητα στη Ρουμανία. Τέλος πάντων ε, υπάρχουν διαφορετικές μειονότητες που αναφέρονται σε 60 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε βασικά, βασικούς τύπους μειονοτήτων. Αυτό το οποίο δεν ε, άκουσα να συζητιέται σε αυτή τη συζήτηση είναι η, η ίση θέση. Δηλαδή, σύμφωνα με την νομοθεσία υπάρχουν οργανισμοί ισότητος που θα έπρεπε να αναλάβουν την, ε, ε, ε, την διάδοση των πολιτικών αυτών και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των σωστών πολιτικών στις διάφορες χώρες. Κατά τη γνώμη λοιπόν είναι περίεργο ότι δεν έχουμε κοιτάξει τι γίνεται με αυτά, στους τους οργανισμούς ισότητος, διότι ε, νομίζω ότι το προσωπικό των οργανισμών αυτών είναι ανεπαρκέστατο σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κατόπιν της εθνικής νομοθεσίας. Είναι 4-5 εκατομμύρια άτομα τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλα τους τα καθήκοντα. Αυτό το οποίο έχω σκεφτεί επί του συγκεκριμένου θέματος. Ε, όλοι είδα ότι όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην έλλειψη στοιχείων. Έχουμε ε, τη, τα δημογραφικά στοιχεία, αλλά ε, υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις. Στη δικιά μου χώρα, παραδείγματο χάρη, 80-90 χιλιάδες άτομα έχουν εντοπιστεί σαν ρομ. Ε, ε, οι υπολογισμοί όμως είναι ότι πρέπει να υπάρχουν 400.000 άτομα και αυτό μπορεί να ισχύσει για όλες τις ομάδες των μεταναστών διότι αν αποφασίσουν ότι καλύτερο θα ήταν να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία ποτέ δεν πρόκειται να δεχθούν ότι ανήκουν σε μειονότητα. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να έχουμε στοιχεία και ίσως με την βοήθεια των ε, ε, γραφείων θα μπορούσαμε ε, να ζητήσουμε από τους οργανισμούς ερεύνης να μας δώσουν στοιχεία σχετικά με αυτό το θέμα. Λοιπόν, πολύ σύντομα αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου και σας παρακαλώ να είστε υπομονετικοί και εύχομαι να επιτύχετε σε αυτό το δύσκολο έργο. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ που μας κάνατε αυτά τα σχόλια διότι έθεσαν στο σωστό πλαίσιο ορισμένες προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν σήμερα το πρωί. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Παρβένοβα που διοργάνωσε τη σημερινή ακρόαση. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική και ε, φυσικά δεν έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Έχει δίκιο η κυρία ε, Μπάουερ. Ε, δεν μπορούμε να δούμε συνολικά τα προβλήματα. Υπάρχουν μετανάστες γυναίκες, γυναίκες ρομ. Πρέπει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις αν θέλουμε να εκπονήσουμε σωστές συστάσεις. Το μόνο κοινό σημείο που εγώ βλέπω ανάμεσα σε όλες αυτές οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες είναι το αντικείμενο της ακρόασης, ε, είναι ότι όταν υφίσταται διάκριση ή καταπίεση μία ομάδα, οι γυναίκες ε, υφίστανται διπλή καταπίεση. Ε, αυτό είναι το κοινό σημείο που μπορούμε να δούμε για τις, ανάμεσα στις μετανάστριες, τις ΡΟΜ κτλ. Και γι' αυτό το λόγο εγώ ασχολήθηκα μόνο με τις γυναίκες Ρώμα και δεν αναφέρθηκα καθόλου στις μετανάστριες, ε, διότι στην περιοχή μου αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί πολύ συχνά. Επίσης, ε, πρόσφατα στις 25 ε, Μαρτίου υιοθετήσαμε μία σύσταση στο Κοινοβούλιο για την δεύτερη Ευρωπαϊκή Σύνοδο για τους δρόμους στην Κόρδοβα και λυπούμε διότι δεν ελήφθηκε όντως υπόψη ε, το θέμα της ισότητας των δύο φύλων ε, παρά, παρόλες τις προσπάθειες που καταβάλαμε εμείς ε, θα πρέπει να καλύψουμε κάποια στιγμή αυτό το χάσμα διότι υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσουμε υπέρ των γυναικών. Η διάκριση λοιπόν που υφίστανται οι γυναίκες ΡΟΜ ε, εντοπίζεται στην άσκηση των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Απασχόληση, υγεία, εκπαίδευση, τα συζητήσαμε όλα αυτά. Τώρα, ε, ε, καταπιέζονται οι γυναίκες ΡΟΜ στον τομέα της υγείας. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες γιατί οι εμπειρογνώμονές μας μας μίλησαν επί μακρόν για αυτό το θέμα και βάσει των γιατρών του κόσμου ε, η πρώτη εγκυμοσύνη έρχεται στα 17 χρόνια. Μόνο 10% των ΡΟΜ έχουν ε, αντισύλληψη. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δεδομένα. Το εκπαιδευτικό σύστημα επίσης αναφέρθηκε. Το θέμα των ειδικών ομάδων, των στα σχολεία ε, των ειδικών τάξεων, δηλαδή τα παιδιά ΡΟΜ, ε, που επειδή είναι ΡΟΜ μπαίνουν στις ίδιες τάξεις με ανάπηρα διανοητικά καθυστερημένα παιδιά, είναι ζητήματα που πρέπει να μα απασχολήσουν. Η πρόσβαση στην απασχόληση τώρα, οι δυσκολίε, ο πιστό, η παρενόχληση, ε, σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, υπάρχουν σημαντικές μαρτυρίες. Γι' αυτό οι γυναίκες σε Ρώμη υφίστανται λοιπόν ε, ε, πολύ ισχυρές διακρίσεις λόγω της εθνοτικής προέλευσης. Ε, χαίρομαι που η Ισπανική Προεδρία της Ένωση. Ε, αναδεικνύει σε προτεραιότητα αυτό το θέμα και ελπίζω ότι από αυτή την πλευρά θα μπορέσουμε τελικά να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν συζητηθεί πρόσφατα ε, εδώ και σε άλλα βήματα. Θα ήθελα εντάχει να αναφέρω κάποιες ιδέες που μπορεί και να ε, συνιστούν λύσεις, γιατί αυτό μας δίσατε να κάνουμε, να προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο. Χρειαζόμαστε μια πολιτική, ειδικά για τις γυναίκες Ρώμα, μια στοχευμένη πολιτική που ως εκ τούτου θα είναι και πιο αποτελεσματική πολιτική, να προβάλλουμε αυτή την πολιτική. Είναι σημαντικό να είναι στοχευμένη η πολιτική. Για την υγεία χρειάζονται ε, εκπαιδευτικά σεμινάρια κατά των προκαταλήψεων για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, ε, κυρίως ε, ως προς τους υπαλλήλους των κρατικών φορέων, γιατί και εντοπίζονται τα βασικότερα προβλήματα. Επίσης, το θέμα της γλώσσας στα νοσοκομεία αντιμετωπίζουμε συχνά αυτό το πρόβλημα, δηλαδή η επικοινωνία ανάμεσα στο προσωπικό των νοσοκομείων και τις γυναίκες Ρώμα η δυσκολία επικοινωνίας που μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση επίσης, χρειάζεται Ε, και μιλώ για κάποια νοσοκομεία ή άλλε δημόσιε υπηρεσίε. χρειάζονται μεταφραστέ, ε, ούτω ώστε να αποφύγουμε ε, πολύ μεγάλα λάθη που γίνονται στον τομέα της υγείας, ε, έχουν κατατεθεί σχετικέ μαρτυρίε, ακόμη και αμβλώσει που δεν επιθυμούν οι γυναίκε, έχουν προκύψει λόγω τη έλλειψη επικοινωνία. Επίση, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το αναφέραμε αυτό, παραβίαση τη σωματική ακαιρεότητά του με υποχρεωτική στήρωση, χαρή, κάποια κράτη-μέλη έχουν αποζημιώσει, έχουν διορθώσει αυτό το πρόβλημα, κάποιε άλλε όχι. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ή υποψήφιε χώρε ε, οπωσδήποτε απαραίτητα θα πρέπει να ρυθμίσουν αυτό το πρόβλημα εφόσον το έχουν αντιμετωπίσει. Το πρόβλημα δηλαδή τη υποχρεωτική στήρωση. Πρέπει οπωσδήποτε να διοργανώσουν επίσημε έρευνε, πλήρει, αμερόληπτε έρευνε για αυτό το φαινόμενο. Οι γυναίκε ε, το χρειάζονται. Πρέπει να αποδοθεί η δικαιοσύνη, να αναγνωριστεί ότι έχουν πέσει θύματα αυτών των πρακτικών και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να προβλεφθούν αποζημιώσει ε, για τα θύματα και οι υπέτειοι ε, να υποστούν κυρώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδοθεί δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βάλλοντε οι γυναίκε Ρώμη επίση ω προ τον κίνδυνο που υπάρχει να πέσουν θύματα εμπορία ανθρώπων και καταναγκαστική πορνεία. Ε, το Κοινοβούλιο στι 14 Ιανουαρίου 2009 εξέδωσε μία σύσταση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρονται οι γυναίκε Ρώμη. Όσα κράτη λοιπόν λοιπόν ε, δεν συμμορφώθηκαν με την νομοθεσία για την καταπολέμηση τη εμπορία ανθρώπων θα πρέπει να δράσουν άμεσα και να συμμορφωθούν. Ε, για το θέμα τη εκπαίδευση ε, το συζητήσαμε ήδη, αλλά όντω είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στα κορίτσια, στι νέε γυναίκε. Είναι στοιχείο κλειδί αυτό για τη χειραφέτησή του. Σε κάποια κρατημέλη είναι τέτοια κατάσταση ώστε να πρέπει να δράσουν οι υπάλληλοι δημόσια διοίκηση, δημόσιοι υπάλληλοι, μιλήσαμε για όσοι έχουν πέσει θύματα επιθέσεων που δεν ε, κάνουν καταγγελίε ε, γιατί ε, δεν τους προστατεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πρέπει να αναβαθμίσουμε την υποδοχή τους σε όλε τι κρατικέ υποδομέ, σε όλε τι κρατικέ υπηρεσίε. Ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν για όλα αυτά τα ζητήματα και πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγουμε ζητήματα όπως ε, ε, ε τους ή τους καταναγκαστικούς γάμους ε, και να εργαστούμε για την πρόληψη. Ένα λεπτάκι για την πέρδεψα και τις σελίδες μου. Συνεχίζω με τις προτάσεις που θέλω να κάνω. Για την ε, ισότητα των δύο φύλων έχω κάποιες πιο συγκεκριμένες προτάσεις να κάνω. Προτείνω, παραδείγματο χάρη, να δημιουργηθεί μία μονάδα ειδική για το, τις γυναίκες ρώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Δύο Φύλων. Εφόσον έχουμε πλέον αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, θα ήταν ενδιαφέρον ε, μία μονάδα, μία υπηρεσία να αφιερωθεί στις γυναίκες των ΡΟΜ εφόσον μιλούσαμε για συλλογή ε, στατιστικών δεδομένων, μπορούμε να δράσουμε μέσω αυτή τη μονάδα. Επίση, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να θεσπιστεί ένα θεσμό ειδικού απεσταλμένου για τι γυναίκε στο Ρώμα, ώστε να υπάρξει οριζόντια ενσωμάτωση σε όλε τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση του ζητήματο του Ρώμα, κυρίω των γυναικών Ρώμα, ούτω ώστε να μπορέσει να υπάρξει έλεγχο και ουσιαστική υλοποίηση των ευρωπαϊκών μέσων που αποσκοπούν στην προστασία των εθνικών μειονοτήτων και συγκεκριμένα των γυναικών. Μια άλλη πρόταση που ε, προκρίνω είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου για τους Ρώμα που διαμένουν στην επικράτεια της Ένωσης. Ένα τέτοιο εργαλείο που θα προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής των Ρώμ ε, θα ε, ήταν ιδιαίτερα υποφελές για τις γυναίκες Ρώμ γιατί έτσι θα αναγνωρίζεται η υπηρετική ηθαγένειά τους, η ευρωπαϊκή τους ηθαγένεια και η ελεύθερη κυκλοφορία στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, και το ανέφεραν και συνάδελφοι, αλλά θέλω να επιμείνω γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Οι οργανώσεις των γυναικών Ρώμα και οι οργανώσεις των Ρώμα γενικότερα, όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ρώμ και των ε, ταξιδιωτών, των διπώνων, θα πρέπει να συνεργαστούν και να εντάσσουν τη δράση τους στη γενικότερη πολιτική της Ένωσης. Ε, για τις γυναίκες Ρώμ και γενικότερα για τους Ρώμ πρέπει οπωσδήποτε ε, οι ευρωπαϊκές πολιτικές να λάβουν υπόψη, παραδείγματος χάρη, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για όλες αυτές τις οργανώσεις. Είναι σημαντικό να συμμετάσχουν αυτές οι οργανώσεις και να συνεργαστούμε εμείς με αυτές τις οργανώσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Κιλ Νίλσεν. Προτείνω τώρα να ακούσουμε την κυρία Παρβάνοβα τώρα, την συγγήτριά μας. Ε, θέλω και εγώ να, με τη σειρά μου να την ευχαριστήσω για τη διοργάνωση της ε, σημερινής ε, ακρόασης. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως το θέμα αυτό είναι ευαίσθητο και δύσκολο και όπως είπε και η κυρία Μπάουερ, ε, μάλλον όχι μόνο εγώ αλλά όλες μας χρειαζόμαστε πάρα πολύ θάρρος και αλληλοϊποστήριξη. Θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε μέχρι στιγμής για εμένα ε, η έλλειψη ορισμού είναι μήνυμα μιας ενιαίας ε, προσέγγισης και μιας ε, πρόθεση και πολιτικής βούλησης για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Και παρά το ότι αυτό δεν είναι εμπόδιο, νομίζω πως σήμερα ακούσαμε την άποψη των ανθρώπων, όπως είπαμε, από τη βάση και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αφού προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πολιτική από πάνω προς τα κάτω, να ξεκινήσουμε με τα μικρά αλλά σημαντικά για τους ανθρώπους στη βάση. Και πιθανότατα έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Σας ευχαριστώ για τις θαυμάσιες ιδέες ε, που ακούσαμε, σημειώσαμε όλα τα προβλήματα και βέβαια στην αρχή ανέφερα κάποια από αυτά, την εκπαίδευση, τη στέγαση, απασχόληση, υγεία. Τώρα έχουμε τη γλώσσα, το θεσμικό πλαίσιο, τη διοίκηση, τη χρηματοδότηση, τη φτώχεια. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που πρέπει να δούμε και από την πλευρά των μειονοτήτων. Βία, σωματεμπορία, πορνεία, καταναγκαστική πορνεία, συλλογή δεδομένων και έρευνα και βέβαια η δίκαιη αντιμετώπιση των μειονοτήτων και η αντιμετώπιση των δικών τους ε, προβλημάτων, ειδικά στο πλαίσιο της ε, οικονομικής κρίσης. Βεβαίως, Υπάρχουν διαφορετικές μειονότητες, διαφορετικές ομάδες, κάποιες είναι εδρεωμένες, ιστορικές αν θέλετε, άλλες ε, είναι αποτελείται από ανθρώπους που ήρθαν πρόσφατα. Υπάρχει και διαφορά στο φύλλο βεβαίω σε κάποιες μειονότητες. Όπως ακούσαμε από κάποιους μειονότητες έρχονται περισσότερες γυναίκες. άλλες μετακινούνται οικογενειακώς ή κατά βάση οι άντρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η διαφορά αυτή πρέπει να μας οδηγήσει σε διαφοροποίηση, στην αντιμετώπιση, στην ανεκτικότητα. Η Ευρώπη είναι για όλους τους πολίτες ε, και πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους και αντιμετώπιση όλων. Όλοι πρέπει να έχουν, το... πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα τουλάχιστον. Γι' αυτό να ξεκινήσουμε με τα σοβαρότερα προβλήματα παρά το ότι έχουμε κυβερνήσεις που είναι ευαίσθητες στον ορισμό της μειονότητας, πιθανώς βεβαίω για ιστορικούς λόγους, αλλά η καταπολέμηση των διακρίσεων και οι ευκαιρίες και η ισότητα των φύλων είναι βασική αξία για όλους μας. Και εάν ξεκινήσουμε από αυτή την προοπτική, θα διηγηθούμε σε καλύτερες λύσεις και με καλύτερο αντίκτυπο και πραγματικά πιστεύω θα έχουμε στις βέλτιστες πρακτικές. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και βασίζομαι στις προτάσεις σας, τα σημειώσαμε όλα και βέβαια θα βασιστώ και στην στήριξή σας όταν θα συζητήσουμε την έκθεση, θα βάλουμε κάθε προσπάθεια να έχουμε μία έκθεση μέχρι τις 16 νομίζω. Απριλίου και βεβαίως ε, είναι πολύ χρήσιμε οι συνεισφορέ σα. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ κυρία Παρβάνοβα για την ε, σύνοψη των όσων σημειώσατε από την σημερινή ακρόαση. Βεβαίως και εγώ θέλω ε, να ευχαριστήσω και να συμφωνήσω με όσους ευχαρίστησαν γιατί βλέπουμε ότι καταρχήν θα πρέπει να βασιστούμε στο, στα ισχύοντα μέσα στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία σαν Επιτροπή Γυναικών και να εξασφαλίσουμε η νομοθεσία αυτή να εφαρμόζεται ουσιαστικά σε όλες τις χώρες μέλη. Ήδη εκεί χρειάζεται να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρό. Επίσης άκουσα από πολλούς να ζητούν στατιστικές αλλά θα πρέπει να εστιαστούμε στα συγκεκριμένα μέτρα διότι διαφορετικά όλοι και όλες σε αυτή την Επιτροπή για την ισότητα των φύλων επιθυμούν τα, τα θέματα ανισοτήτων να ληφθούν υπόψη και να επιληθούν. Ε, σύμφωνο με την ε, μέθοδο που χρησιμοποιήσατε ε, και που μου φαίνεται πολύ βασική, σημείωσα την συσσόρευση των προβλημάτων ε, κοινωνικών ανισοτήτων σε, στα ίδια άτομα και είδαμε σήμερα το πρωί άλλωστε ότι ε, ε, ο αλφαβητισμός και η πληροφόρηση είναι τα κλειδιά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επίλυση άλλων προβλημάτων όπως η υγεία, η ένταξη. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλες που, και όλους που ήρθαν να περάσουν το πρωινό μαζί μας. Ευχαριστώ και τους, ε, τους βουλευτές. Ευχαριστώ και εύχομαι κουράγιο στην κυρία Παρβάνοβα. Θέλω να ευχαριστήσω και την γραμματεία της Επιτροπής και όλους τους διερμηνείς οι οποίοι μας συνόδευσαν και που επέτρεψαν εις